Προτείνω να αρχίσουμε τη συνεδρίαση, σημείο 1, έγκριση. Μπορούμε να εγκρίνουμε χωρίς τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη, έχετε παρατηρήσεις, εγκρίνεται. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Σας καλωσορίζω. Ελπίζω να περάσατε ωραίες διακοπές. Όπως ε, θα παρακολουθήσατε τις τελευταίες μέρες, η κατάσταση στη Λιβύη εξελίχθηκε σημαντικά. Οι Λίβοι επαναστάτες ελέγχουν ε, σχεδόν ολόκληρη την πρωτεύουσα. Το καθεστώς του Καντάφη έχει πέσει, αλλά ο Καντάφη αγνοείται και παραμένει επιβλαβής. Η συνεδρίαση για την υποστήριξη της Λιβύης θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου στο Παρίσι. Θα γίνει μία ανταλλαγή απόψεων με τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την περιοχή, τον κύριο Λεόν. Σήμερα το απόγευμα θα τον ακούσουμε. Θα μιλήσουμε για τη Λιβύη αλλά και για τη Συρία. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να εγγραφείτε για τις τοποθετήσεις σας στην ακρόαση με τον κύριο Λεόν σήμερα το απόγευμα. Σημείο 3. Πρακτικά 24η-25η Μαΐου, 6 Ιουνίου, 15-16 Ιουνίου, 21 Ιουνίου, 27 Ιουνίου. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, εγκρίνονται. Και πάμε τώρα στο σημείο 4, το στάδιο εφαρμογής της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία. έκθεση της κυρίας Κιλ Νίλσεν για την εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία που περιλαμβάνει χώρες με ιδιαίτερα στρατηγική σημασία με μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες, αλλά που έχουν σημαντικά προβλήματα σε, στον τομέα της σύγκλησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τον Απρίλιο η Επιτροπή μας ακροάστηκε εδώ ε, υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου πριν από την επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στις χώρες της περιοχής. Ουζουμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν. Το Μάιο οργανώσαμε μία ακρόαση εμπειρογνωμόνων για την γεωστρατηγική της ενέργειας, του ύδατος και του κράτους δικαίου. Όλα αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν στη σύνταξη της, κυρί... της έκθεσης της κυρίας Νίλσεν και δίνω την, το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Κιλ Νίλσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως ε, όλοι το γνωρίζετε από το 2007 και μετά ξεκίνησε μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται. Όπως το λέω και στο αιτιολογικό που σίγουρα το διαβάσατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε πρωτοβουλίες και δεν θα επανέλθω σε αυτά, διότι εκτίμησα ότι θα ήταν χρήσιμο να συνταχθεί αυτή η νέα έκθεση, διότι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να επανέλθουμε στη στρατηγική μας αυτή την περιοχή, και αυτό λόγω των ορίων αυτών των στρατηγικών, τα οποία πλέον έχουμε αρχίσει και διαπιστώνουμε, αλλά και λόγω των νέων αλλαγών, τόσο παγκοσμίως όσο και στις περιοχές αυτές. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, η έκθεση αφορά στη δική μας στρατηγική για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι μια έκθεση που αφορά τις χώρες αυτές. Η στρατηγική μας έχει ορίσει 7 βασικές προτεραιότητες στο αρχικό της έγγραφο, να σας τις θυμίσω. Εκδημοκρατισμό, εκκυβερνησία, εκπαίδευση, οικονομία, εμπόριο, ενέργεια, μεταφορές, περιβάλλον, διαχείριση του ύδατος, καταπολέμηση των απειλών και των κοινών προκλήσεων, πολιτιστική συνεργασία. Καταλαβαίνετε ότι στην έκθεσή μου δεν μπορεί κανείς να εξετάσει όλα αυτά τα σημεία. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι να δούμε ποιες είναι οι πιο πιεστικές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι σημαντικό να εργαστούμε για τα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ενέργεια, την περιφερειακή ασφάλεια. Αυτά τα σημεία τα εξετάζουμε ως εξής. Έχουμε δύο πυλώνες, ανθρώπινη ασφάλεια και περιφερειακή συνεργασία. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί πυλώνες. Έτσι εγώ διαρθρώνω την έκθεσή μου. Ανθρώπινη ασφάλεια θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι θα πρέπει η η αιρεσιμότητα να αποτελεί απαράβατο όρο για τις πολιτικές μας, όχι μόνο σε αυτή την περιοχή αλλά και αλλού. Βλέπετε τι γίνεται στις αραβικές χώρες και όλα όσα διαμείβονται εκεί θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε σκέψη για τη στρατηγική μας στην Κεντρική Ασία, για τις προτεραιότητές μας και τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει να εργαστούμε. Ανθρώπινη ασφάλεια λοιπόν. Δεύτερο, περιφερειακή συνεργασία είναι ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό. Όλες οι προκλήσεις στην περιοχή, δηλαδή διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο όπλων, λαθρεμπόριο όπλων, το νερό, διαχείριση των φυσικών πόρων κλπ. Όλα αυτά δεν μπορούν να επιληθούν χωρίς διαβούλευση με τις ε, χώρες της περιοχής. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο και το διαπιστώνω και το διαπιστώσαμε ότι οι χώρες της Κεντρικής Ασίας παρά ορισμένα επιχειρήματα και λοιπά δεν είναι και τόσο διαθέσιμες για συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ουδέτερη είναι και την ιστορική εμπειρία έχει, οπότε έχει και τη δυνατότητα να σμπρώξει τα πράγματα. Αυτό δεν αντιφάσκει με αυτό το οποίο λέγεται στην έκθεση, ότι θα πρέπει να έχουμε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση έναντι των πέντε χωρών. Δεν είναι, έλεγα, αντιφατικό. Πρέπει να έχουμε μια διαφοροποιημένη διμερή προσέγγιση ανάλογα με την ανάγκη της κάθε χώρας. Είναι η πρώτη παρουσίαση της έκθεσής μου και είναι σημαντικό καθένας από εσά να εκφραστεί και να υποβάλει προτάσεις. Εγώ περιμένω συνεργασία από τους συναδέλφους και ελπίζω να έχω προτάσεις από τον καθένα σας. Αυτό το οποίο θα ήθελα ήταν να, να σας δώσω το βασικό πλαίσιο της έκθεσης. Υπάρχουν μερικά μεταφραστικά λάθη στην γαλλική έκθεση, στην παράγραφο 3. Είναι σημαντικό σημαντικό να πούμε ότι δεν δεν αναθέτουμε στις μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ, αλλά καλούμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να συμμετέχουν. Υπάρχει και ένα λάθος για το Ουζουμπεκιστάν, η άρση των κυρώσεων για το Ουζουμπεκιστάν. Ουζουμπεκιστάν λαμβάνει υπόψη τις ε, αποφάσεις του Συμβουλίου του 2008 και όχι του 2010. Αυτά σας τα λέω για να τα ξέρετε να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Για τα θέματα της ασφάλειας, της ανθρώπινης ασφάλειας, ε, υποβάλλω προτάσεις και έχουμε ε, την πρόταση για το φόρουμ, το κοινοβουλευτικό φόρουμ, να παίξουμε δηλαδή ένα ρόλο ε, κινήτρου έλκυσης για να προχωρήσει η ίδια περιφερειακή συνεργασία. Για το θέμα της ανθρώπινης ασφάλειας θέλω να σας διευκρινίσω ότι η παράγραφοι και αυτό λόγω διακοπών, μεταφράσεων κλπ. η παράγραφοι έλεγα έχουν προσθεθεί από μένα εκ των υστέρων, δεν βρίσκονται δηλαδή στο έγγραφο. Πρόκειται για μια πρώτη απάντηση που δίνω εγώ στο πρόβλημα, προσδοκώ πολλά από τους συναδέλφους για να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Σημειώσαμε. όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, υπομορφή διορθώσεων. Θα ήθελα να στραφώ τώρα στους συζητητές για το ΕΡΚ. Η κυρία Βέτερε ε, αντικαθιστά την κυρία Σίγκολ, η οποία είναι σκιώδη εισηγήτρια για το θέμα αυτό. Έχετε λοιπόν, κυρία Ντεβέντερε, το λόγο. Good morning, dear colleagues. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως πληροφορηθήκατε, πρέπει και εγώ να σας πω ότι η κυρία Γέγκλε είναι σε μια επίσημη αντιπροσωπεία και δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα. Εγώ θα μιλήσω εξ ονοματό τη. θα παρουσιάσω τα κύρια θέματα στη σχέση με αυτό το σχέδιο έκθεση και θα ήθελα επίση να σα αναφέρω ότι όχι μονάχα αντικαθιστώ την κυρία Γέγκλε, αλλά θέλω να εκφράσω και τι δικές μου απόψει γιατί συμφωνούμε σε όλα τα σημεία με την κυρία Γέγκλε. Και εγώ ταξίδευσα στις χώρες της Κεντρικής Ασίας πολλές φορές. Ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση εκεί. Και φυσικά πρέπει να ευχαριστήσω καταρχήν την κυρία Κιλ Νίλσεν για το σχέδιο εκθεσή τη και για τι προσπάθειε που κατέβαλε σε σχέση με τις χώρες κεντρική Ασίας παρά τι διακοπέ. Γιατί πρέπει να έχουμε μια έκθεση λοιπόν για τι χώρε αυτέ. Πρέπει καταρχήν να υπογραμμίσουμε τη σημασία που επέχουν οι χώρε αυτέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τούμπαλιν και πρέπει να εξηγήσουμε του λόγου για του οποίου είναι απαραίτητη η συνεργασία μα είναι όμορες χώρες προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από γεωγραφική έποψη. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξασφαλίσουμε τη σωστή διακυβέρνηση, το κράτο δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία κτλ. Η κυρία Γέγλε ήθελε να υπογραμμίσει ιδιαίτερα και εγώ το ίδιο ότι η οικονομική ανάπτυξη και η δημοκρατία, ο εκδημοκρατισμό είναι αλληλένδετες έννοιες και συμπληρωματικού χαρακτήρα. Οι χώρες αυτές έχουν να αντιμετωπίσουν ε, θρησκευτική ακεροφροσύνη λόγω και της εγκύτητό τους στο Αφγανιστάν. Δεν πρέπει λοιπόν να παραμερίσουμε τις περιοχές αυτές. Χρειάζεται μια βιώσιμη και συνεχής συνεργασία με τις χώρες αυτές. Μερικά ακόμα κομβικά σημεία τα οποία αναφέρονται στο σχέδιο της κυρίας Κιλ Νίλσεν. Εμείς συμμεριζόμαστε την άποψη αυτή ότι μια ορατή παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, στις χώρες αυτές είναι απαραίτητη. Είναι πολύ σημαντική και η παρουσία μας με τις αντιπροσωπείες και τα λοιπά και υποστηρίζουμε την ιδέα του να υπάρξει μια σειρά από κοινοβουλευτικέ επαφέ μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρών τη Κεντρική Ασία. Είμαστε πεπισμένοι επίση ότι η συνεργασία στα θέματα διαχείριση υδάτινων πόρων με τι χώρε αυτέ είναι κάτι το οποίο είναι απαράγραπτο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένα διαμεσολαβητή για την καλύτερη χρήση αυτών των πόρων. Ένα άλλο σημείο το οποίο θέλουμε να προσθέσουμε στο σχέδιο έκθεσης είναι το εξής. Προτείνει η κυρία Γέγλε να υπάρξει και ένα κεφάλαιο για οικονομική ανάπτυξη που να περιλαμβάνει και την υποστήριξη σε μια ενισχυμένη οικονομική συνεργασία στο νέο πλαίσιο που αναδύεται σε παγκόσμιο επίπεδο για να μειωθεί η η ένδια και να ανέλθει το βιωτικό επίπεδο. Επίσης αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον πολλαπλασιασμό των εμπορικών εταίρων για τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, συνεργασία σε προγράμματα υποδομής, προετοιμασία ενός περιβάλλοντος που να είναι φιλικό προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως να εξάρουμε και να ενισχύσουμε το ρόλο των γυναικών και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μια πιο υποφελή σχέση. <clears throat> Θέλουμε να υπάρξει μια εντατικοποίηση της συνεργασίας σε σχέδια ε, παιδείας με ανταλλαγή διδασκόντων και διδασκομένων και επίσης η κυρία Γέγλε υποστηρίζει το έργο των πολιτικών ιδρυμάτων διότι δημιουργούν και μεταλαμβαδεύουν μακροχρόνια πολιτική εμπειρία στις χώρες αυτές. Κατά την άποψή μας, κυβερνήσεις των χωρών της Κεντρικής Ασίας θα πρέπει να προχωρήσουν στην στεναρή εφαρμογή πολιτικών εγχειρημάτων σε σχέση με τη δημοκρατικοποίηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθήσει από πολύ κοντά τα εγχειρήματα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ακόμα και μικρά βήματα είναι πάντα θετικά. Τέλος, η υπομορφή κατακλείδος, εμείς αναγνωρίζουμε πλήρως το γεγονός ότι η διαδικασία εκδημοκρατισμού και κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης στην Κεντρική Ασία είναι μόνο στα γενοφάσκια της. Επομένως έχουμε πολύ δρόμο να διατρέξουμε. Η πρόοδος στους χώρους αυτούς δεν είναι άμεσα συγκρίσιμη με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και μικρά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση θα πρέπει να τύχουν τις επιδοκιμασίες μας. Είναι λοιπόν μεγάλη σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί και να εμπλακεί ενεργά στην περιοχή αυτή. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε περαιτέρω ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σβόμποντα ως ε, εισηγητής, ε, σκιώδης εισηγητής για τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας την εισηγήτρια για το έργο το οποίο έφερε σε πέρας και την ε, σοβαρότητα της έκθεσής της. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε μερικά θέματα τα οποία ίσως θα έπρεπε να τονιστούν περισσότερο στην έκθεση. Αυτό δεν αποτελεί επίκριση, απλώς θα ήταν η θέλησή μας να υπάρξει μεγαλύτερη έμφαση. Προφανώς δεν πρόκειται για μια έκθεση για τη σύνολη περιοχή, αλλά για την ευρωπαϊκή στρατηγική έναντι της περιοχής της Κεντρικής Ασίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι σαφές. <clears throat> Έχουμε πολλαπλό ενδιαφέρον για αυτή την περιοχή και φυσικά αυτή είναι μια έκθεση η οποία δεν πρόκειται να διαβαστεί από όλο τον πληθυσμό, αλλά θα ήταν χρήσιμο να εξηγήσουμε σε εισαγωγικό επίπεδο γιατί μας ενδιαφέρει αυτή η περιοχή. Παραδείγματο χάρη τα θέματα ενέργειας. Έχουμε προφανώς ένα ενδιαφέρον για του ενεργειακού πόρους για να εξασφαλίσουμε και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής αυτής. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι δύο μεγάλοι, άλλες δύο μεγάλες πολιτικές οντότητες, η Κίνα και η Ρωσία που ενδιαφέρονται για αυτή την περιοχή. Αν εμείς δεν δράσουμε με τρόπο αποφασιστικό μπορεί να βρεθούμε στο περιθώριο και να αφήσουμε αυτή την περιοχή να περιέλθει στην ε, σφαίρα ενδιαφέροντος αυτών των μεγάλων δυνάμεων. Τα θέματα ασφαλείας επίσης είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι αυτή η περιοχή ή τουλάχιστον ορισμένε από τις χώρες αυτές της περιοχής βρίσκονται πολύ κοντά στο Αφγανιστάν. Και επομένως μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η τουλαχιστον ορισμενε απο τι χωρε αυτες τη περιοχη βρισκονται πολυ κοντα στο αφγανισταν και επομενω μας ενδιαφερει ιδιαιτερα η επιτευξη της ε, σταθερότητα στην περιοχή αυτή και δεν θέλουμε να επηρεαστεί από πολεμικές ενέργειες στο Αφγανιστάν και σε άλλε χώρε. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε μια συνεργασία και σε θέματα ασφάλεια με την περιοχή αυτή. Ένα άλλο θέμα είναι η... και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Γνωρίζουμε ότι πολλέ από τι ροέ ναρκωτικών μπορεί να διέρχονται από τι χώρε αυτέ, Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε τον έλεγχο λοιπόν των ροών ναρκωτικών και αυτό μπορεί να γίνει μονάχα με συνεργασία με τι χώρε αυτέ, όχι μόνο προφανώ με αυτέ τι χώρε, αλλά σίγουρα εμπλέκοντα και τι χώρε αυτέ. Όλα αυτά είναι κάποια σημεία τα οποία για μα από τη δική μας πολιτική ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να υπογραφούν, να υπογραμμιστούν. Και φυσικά πρέπει να τονίσουμε και το ενδιαφέρον μας για την πορεία προς τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρόοδος προς την ε, δημοκρατία έχει δίκιο η προλαλή σα, αν δεν μπορούμε προφανώ να συγκρίνουμε τι χώρε αυτέ με τι ευρωπαϊκέ χώρε, οι οποίε έχουν τελείω διαφορετικέ παραδόσει για τα θέματα τη δημοκρατία. Αλλά τονίζω και εγώ ότι χωρί πρόοδο στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούμε να επιτύχουμε μια λογική πολιτική σταθερότητα και μια κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή αυτή. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίζουμε πάντα το θέμα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε δει και στο παρελθόν ότι ο διάλογος δεν είναι εύκολος, <clears throat> αλλά ε, είδαμε ότι δεν είναι αδύνατο να υπάρξει πρόοδος στην περίπτωση του Ουσβεκιστάν, στο Τουρκουμενιστάν επίσης είχαμε πολλές δυσκολίες και είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε και σε περαιτέρω πρωτοβουλίες. Αυτό έδειξε και η επίσκεψή μας στις χώρες αυτές. Πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο μας να δείξει το ενδιαφέρον του και την προσήλωσή του να υπάρξει μια μόνιμη στρατηγική έναντι των χωρών αυτών. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σε χώρες όπως το Καζακστάν, ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες αυτές. Έχουμε λοιπόν επίσης και ένα νέο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και προφανώς είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε σε αυτό το νέο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη δυνατότητα να έρθει ενώπιον της Επιτροπής μας και να ακούσουμε τις απόψεις του και τονίζω το πόσο σημαντική λοιπόν η έκθεση κυρία κυρίας Κίρνιτσεν και η περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Ένα ακόμα σημαντικό σημείο το οποίο θέλω να αναφέρω είναι το σημείο 18. Εδώ αναφέρεται το θέμα της συμμετοχής του Καζακστάν στην Τελωνιακή Ένωση με τη Λευκορωσία και την Ρωσία. Αυτό φυσικά δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε. Αυτό είναι μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί από την ίδια τη χώρα αυτή, το Καζακστάν. Ξέρω ότι υπάρχουν και πιέσεις προς την Ουκρανία να συμμετάσχει σε αυτή την τελωνιακή ένωση, κάτι το οποίο θα δυσκολεύσει ενδεχομένως τις σχέσεις της χώρας αυτής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε λοιπόν αυτή την πορεία προς την Τελωνιακή Ένωση. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να δούμε και τις θετικές πτυχές οι οποίες μπορούν να προκύψουν από μια τέτοια συμφωνία, διότι ευνοούν την περιφερειακή συνεργασία. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν μια κριτική στάση για την Τελωνιακή Ένωση, αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και γι' αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε αυτό που είπε και η κυρία Κίλ Νίλσεν, ότι η πολιτική φιλοσοφία των ηγετών των χωρών αυτών απέχει αρκετά από την φιλοσοφία την πολιτική της ε, Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο και όχι με τους μεγάλους γείτονες των χωρών αυτών. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ε, θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες προς την κατεύθυνση στο σημείο που προανέφερα. Ευχαριστούμε. Κύριε Νικολάη, θέλετε κι εσείς το λόγο εκ μέρους των φιλελεύθερων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Με τη σειρά μου θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και όλα τα προβλήματα τα οποία θίγει στα πλαίσια της έκθεσής της. Και επίσης θέλω να τη συγχαρώ για τον τρόπο με τον οποίο έχει ετοιμάσει την αιτιολογική της έκθεση. Όμως η γενική κατεύθυνση της έκθεσης αυτής, κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να υπογραμμίζει περισσότερο τη συνεργασία με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και την συνεργασία των χωρών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια στην περιοχή. Το κύριο πρόβλημα έχει να κάνει με τον ίδιο τον τίτλο της έκθεσης κατά τη γνώμη μου, γιατί μιλάμε για το στάδιο εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία, ενώ στην έκθεση μιλάμε περισσότερο εξειδικευμένα για την κάθε χώρα. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ και τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Πρέπει να φανούμε αντικειμενικοί. Ο κύριος στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη συνεργασία. Φυσικά και πρέπει να υπογραμμίσουμε τα προβλήματα που παραμένουν στην περιοχή, να τα θίξουμε, να τα επικρίνουμε, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι η κριτική μας αυτή πρέπει να γίνει από την πλευρά ενός ουδέτερου παρατηρητή. Δεν πρέπει εμείς να δείξουμε ότι δίνουμε μαθήματα στους άλλους. Για τελειώς όσα προσπαθούμε να κάνουμε θα παραμείνουν νεκρό γράμμα και θα είναι μόνο κάποια έγγραφα ή εκθέσεις μας που κανείς δεν θα διαβάσει. Χρειαζόμαστε μία διατύπωση λοιπόν πιο επικοδομητική κατά τη γνώμη μου. Επιπλέον στο έγγραφο αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε περισσότερο ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια πραγματική στρατηγική και όχι μόνο ένα κατάλογο ευσεβών πόθων που περιμένουμε να θέσουν σε εφαρμογή οι χώρες αυτές. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας, κάτι το οποίο δεν γίνεται στην έκθεση αυτή. Το σημείο 1, για παράδειγμα, πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να περιμένουμε εμείς ότι θα αλλάξουν όλα εν μία ανοιχτή στην περιοχή. Όσον αφορά τα σημεία 4 και 6 τώρα, εδώ ναι, συμφωνώ, χαίρομαι που συμπεριλαμβάνονται, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε ακόμα περισσότερο με την περιοχή, ε, δημιουργώντας κάποιες αντιπροσωπείες μας εκεί. Έτσι θα ενισχυθεί ο διάλογος και ο κοινοβουλευτικός, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό. Πρέπει επίσης να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά τι μπορούμε εμείς από την πλευρά μας να προσφέρουμε στους ασιάτες εταίρους μας. Λυπάμαι που δεν αναφέρονται καθόλου εμπορικές συναλλαγές ή οικονομική συνεργασία. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια είναι και αυτά πολύ σημαντικά. Η δικιά μας ενεργειακή στρατηγική πρέπει να λαμβάνει υπόψη το τι συμβαίνει στην περιοχή. Έρχομαι τώρα στο σημείο 11. Όλα όσα αναφέρονται εδώ είναι καλά, αλλά Μιλάμε εδώ πολύ περισσότερο για το περιβάλλον παρά για την ενέργεια. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν θέλουμε η Κεντρική Ασία να πλησιάσει περισσότερο τις ευρωπαϊκές αξίες, τότε οφείλουμε εμείς να ασχοληθούμε περισσότερο μαζί τους. Πρέπει να βρούμε τη δύναμη, πρέπει να βρούμε την αποφασιστικότητα, να το κάνουμε, να είμαστε παρόντες και σε αυτή την περιοχή. Το κεφάλαιο τώρα που αναφέρεται στην ασφάλεια στην περιοχή πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο. Πρέπει να μιλάμε εκεί και για την Κασπία θάλασσα και να μην ξεχάσουμε τι εντάσεις υπάρχουν στην περιοχή ακριβώς εξαιτίας ε, περιφερειακών διανέξεων. Νομίζω ότι το κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται χωριστά σε κάθε μία χώρα δεν ε, έχει παντού ίδιο βάρο. Στο σημείο 25 μου φαίνεται επικοδομητικό, αλλά αυτά που λέγονται εκεί ισχύουν και για τις άλλες χώρες της περιοχής. Και όχι μόνο για τα ενεργειακά προγράμματα, αλλά και για το κοινωνικό τομέα, για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ. κλπ. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μία στρατηγική η οποία ξεκάθαρα να αναφέρει τα όρια της εμπλοκής μας στην περιοχή. Είμαι πεπισμένη ότι τη απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, όλοι οι ευγενείς στόχοι μας θα παραμείνουν απλώς ωραία λόγια. Και βρισκόμαστε σε μια στιγμή της ιστορίας που δεν μπορούμε πια να επιτρέπουμε στους εαυτούς μας τέτοιου είδους συμπεριφορές. Θα υποβάλουμε τροπολογίες και είμαστε πεπισμένοι ότι θα καταλήξουμε σε μία έκθεση η οποία να δείχνει ποια πραγματικά είναι η άποψη και το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Ευχαριστούμε κυρία Νικολάη, πρόεδρος. Σταματάμε εδώ με τους σκιώδεις συζητητές γιατί δεν βλέπω εδώ τον κύριο Τάνοκ από το ΣΥΕΡ. Τώρα περνάμε σε ανταλλαγή απόψεων με τους ευρωβουλευτές. Ο κύριος Σίβικ πρώτα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, Νομίζω ότι η πολιτική θυμίζει μερικές φορές τον αθλητισμό. Νομίζω ότι αυτή η συγκεκριμένη έκθεση μας έρχεται μια πολύ σημαντική και καλή στιγμή. Και λέω ότι είναι μια καλή στιγμή γιατί πραγματικά πρέπει τώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε γενικότερα την ευρωπαϊκή πολιτική. Επίσης είναι μια καλή στιγμή γιατί εγώ είμαι υπεύθυνο για μια άλλη έκθεση που έχει να κάνει με την πολιτική γετνίαση. Και μέχρι τώρα είχα διάφορες επαφές και συναντήσεις και το συμπέρασμα είναι πολύ, πολύ σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη δημοκρατία, να ασχοληθούμε με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία αποτελούν και τη βάση όχι μόνο στο κάτω-κάτω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων χωρών. Πρέπει να παίρνουμε μαθήματα εξάλλου από τα όσα συμβαίνουν στη Βόρεια Αφρική. Χωρίς δημοκρατία, χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα, κάθε άλλο είδους δημοκρατία δεν είναι παρά μεταβατική. Δεν κρατάει δηλαδή στο χρόνο. Τώρα για να επανέλθω στην έκθεση. Οι πέντε χώρες οι οποίες αναφέρονται εδώ μοιάζουν μεταξύ τους με την έννοια ότι μέχρι τώρα έχουν αγνοηθεί πολλά πράγματα σε όλες αυτές τις χώρες, κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει, να γίνουν μεταρρυθμίσεις δηλαδή. Ο παλιός τρόπος που λέγαμε ότι ε, εντάξει όσο είναι ειρηνική η κατάσταση στην περιοχή σας, εμείς θα συνεχίσουμε να σας ανισχύουμε όπως κάνουμε μέχρι τώρα. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις δεν ισχύουν πια. Πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θέλουμε να ενισχύσουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την εκπαίδευση, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τα συστήματα δικαιοσύνης εκεί. Να δούμε πώς θα στηρίξουμε τις κοινωνικές οργανώσεις, πώς αυτές λειτουργούν εκεί. Οπότε τι κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε έκκληση και να διασφαλίσουμε ότι η περιοχή είναι ένας χώρος όπου ισχύει μια συνεκτική πολιτική. Μια τέτοια πολιτική εφαρμόζουμε. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να φτιάξουμε μια πολιτική γετνίαση και για αυτή την περιοχή, αλλά να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε αν μη τι άλλο να δούμε και να εντοπίσουμε τι κοινό υπάρχει μεταξύ των χωρών αυτών. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει αυτό η συγγήτρια. Εμείς πάντως θα υποβάλουμε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου, αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική περιοχή του κόσμου. Υπάρχει η ευρωπαϊκή πολιτική, η πολιτική της Κίνας ή της Ρωσίας στην περιοχή. Υπάρχουν αυτές οι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές πολιτικές. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η περιοχή. Απ' την άλλη δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια επειδή είναι σημαντική η περιοχή και να αφήνουμε μερικά πράγματα χωρίς να τα φύγουμε καθόλου. Κάτι άλλο τώρα από πιο τεχνική άποψη. Η συγκίτρια αναφέρεται εξατομικευμένα στις διάφορες χώρες και καταλήγει σε συμπεράσματα τα οποία είναι σωστά, δικαιολογούνται, αλλά μερικές φορές μου φαίνονται επιφανειακά. Και εγώ, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, έχουμε δουλέψει πάνω σε εκθέσεις για το Τουρκμενιστάν. Και εκεί ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ συγκεκριμένη, πολύ διαφορετική στο Τουρκμενιστάν. Έχουμε επαφές με διάφορες ε, οργανώσεις για να ετοιμάσουμε τις εκθέσεις μας αυτές. Οπότε ίσως αντί απλώς να αναφέρουμε εδώ πέρα διάφορα πράγματα έτσι κοινότυπα που έχουν να κάνουν με τις πέντε χώρες, ίσως να μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας τις εκθέσεις που ετοιμάζουμε για κάθε μία από τις χώρες αυτές και έτσι να καταλήξουμε σε πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πίτερ λέει έχει τώρα το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και κυρίως την εισηγήτρια, την κυρία Νίλσεν, για την ε, τόσο ξεκάθαρη θέση την οποία υιοθετεί και η οποία βασίζεται σε μια πολύ καλή ανάλυση της κατάστασης στην Κεντρική Ασία. Έχω πολιτικές εμπειρίες εγώ προσωπικά από την περιοχή και γι' αυτό πιστεύω ότι έχει στρατηγική σημασία η Κεντρική Ασία. Οι χώρες ε, εκεί μερικές φορές δεν νιώθουν την ανάγκη να συνεργαστούν μεταξύ τους αυτό που τις χαρακτηρίζει είναι ότι η μεταπολίτευση μετά από την ανεξαρτησία τους από τη Σοβιετική Ένωση δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερο, σε ορισμένες λιγότερο και μερικές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Εγώ συμφωνώ πάντως και με την εισηγήτρια και με άλλους ομιλητές για το ότι πρέπει να αγωνιστούμε μέσα σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο για σταθερότητα στην περιοχή. Κατά τη γνώμη μου, εσωτερικά προβλήματα στις χώρες της Κεντρικής Ασίας μπορεί να συνεχίσουν να είναι δύσκολα και να γίνουν ακόμα πιο δύσκολα από ό,τι στη Βόρεια Αφρική. Κάτι στο οποίο αναφέρθηκε προλαλή σας. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώς και πρέπει να δείξει ότι ενδιαφέρεται για τις δημοκρατικές αλλαγές από στρατηγική άποψη στην περιοχή. Πρέπει να αποφύγουμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Εγώ πιστεύω ότι μετά από τέσσερα χρόνια πρέπει να αξιολογήσουμε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή αυτή και χαίρομαι που στην έκθεση υπογραμμίζεται αυτό. Πιστεύω επίσης ότι είναι αναγκαίο να έχουμε αντιπροσωπείες σε όλες τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Με το κατάλληλο προσωπικό, επαρκές κλπ. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω είναι κάτι για την πρόταση να υπάρξει ένα κοινοβουλευτικό φόρουμ με τις χώρες αυτές. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Είναι δικιά μας πρωτοβουλία, έρχεται αποκλειστικά από τη δικιά μας την πλευρά ή το έχουμε ελέγξει κάπως και με τα κοινοβούλια των χωρών αυτών και το υποστηρίζουν και εκείνες. Εγώ προσωπικά γνωρίζω ότι ο διάλογος έχει μεγάλη σημασία και σίγουρα στηρίζω την πρωτοβουλία αυτή, ένα τέτοιο φόρουμ δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πίτερλε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η κυρία Κιλ Νίλσεν έχει συντάξει μια έκθεση η οποία είναι πολύ σημαντική, θετική για την ουσία της και <clears throat> έρχεται σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή. Για τη στρατηγική μας τώρα σε σχέση με την Κεντρική Ασία, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Σφόμποτα ότι πρώτα απ' όλα είναι απαραίτητο να παρουσιάσουμε τους λόγους του ενδιαφέροντός μας σε αυτή την γεωγραφική περιοχή, τα στρατηγικά επιχειρήματα, τα επιχειρήματα ασφάλειας, τα επιχειρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τροφοδοσία σε ενέργεια. Σε ό,τι αφορά την παροχή πετρελαίου και φυσικού αερίου, η έκθεση δεν διαλαμβάνει τα θέματα αυτά περισσότερο αναφέρεται σε υδάτινους πόρους, σε γεωργία κτλ. Νομίζω όμως πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα θέματα της ενέργειας. Επίσης, <clears throat> ένα άλλο θέμα το οποίο αναφέρθηκε από τους προλαλήσαντες είναι οι σχέσεις των χωρών αυτών με το Αφγανιστάν. Εάν όλα πάνε καλά, το Αφγανιστάν θα μπορέσει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο όχι μονάχα από στρατηγική έποψη αλλά οικονομικά και κοινωνικά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των χωρών της σύνολης αυτής της περιοχής. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν και αυτό το θέμα. <clears throat> Επίσης, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλους διεθνείς παίκτες όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και εδώ εμπλέκονται ιδιαίτερα σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή αυτή. Και η Κίνα και η Ρωσία διεκδικούν την επιρροή στην περιοχή αυτή. Επομένω, πρέπει να έχουμε κάποια στρατηγική για το πώ θα αντιμετωπίσουμε συνολικά την περιοχή αυτή και ποιε είναι οι δυνατότητε συντονισμού που ανοίγονται μπροστά μα. <clears throat> Νομίζω ότι και η Γερμανία, καθώ και η Γαλλία, έχουν δώσει το καλό παράδειγμα στα θέματα αυτά και έχουν δώσει σημαντικές συνεισφορές με τις πρωτοβουλίες τους για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά τα οποία υπάρχουν στην περιφερειακή ασφάλεια στην περιοχή αυτή. Η συγγήτριά μας επίσης έχει παρουσιάσει πολύ ορθά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ε, προσέγγιση μας στο σημείο 21 όταν είπε ότι η οικονομική συνεργασία θα πρέπει να προχωρήσει χέρι-χέρι με την πολιτική συνεργασία και με την πολιτική θέληση να εδρεωθούν και να υλοποιηθούν οι κοινέ αξίες μας. Επίσης, το σημείο 29, την παράγραφο 29, εκφράζουμε τη λύπη μας για το κλείσιμο του γραφείου της Human Rights Watch στην Τασκένδη. Νομίζω πρέπει να το πούμε λιγάκι πιο εμφατικά αυτό το θέμα. Να το τονίσουμε λοιπόν. Αλλά εν γέννη συμφωνώ και πάλι για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει την πλήρη της προσήλωση, την πραγματική της προσήλωση για αυτή την περιοχή μας ενδιαφέρει για πολλαπλούς λόγους αυτή η περιοχή και πρέπει να υπάρξει και μια συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού, της εδραίωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περιοχή αυτή. Είναι αποφασιστική λοιπόν στον τομέα αυτό η δική μας δράση, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι διεθνείς εταίροι και παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο εκτός από εμάς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κέλλαμ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φρελέσεν από την Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε <clears throat> και εμείς ε, χαιρετίζουμε το σχέδιο ψήφισματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντρική Ασία. Είναι μια πάρα πολύ εύστοχη και επίκαιρη συνεισφορά η οποία θα συμβάλλει στη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής στο Συμβουλίο μετά από την έγκριση τη Στρατηγική για την Κεντρική Ασία από το Συμβούλιο το 2007 έχουν υπάρξει πολλέ εξελίξει στι σχέσει μα με την περιοχή αυτή. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί στην αξιολόγηση τη στρατηγική μα, Δεν πρόκειται για χώρε οι οποίε είναι υποψήφίε για ένταξη μέσα στην πολιτική γειτονία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. όπου μπορούμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση με του περιορισμένου πόρου τη έχει παίξει σημαντικό ρόλο και μπορεί να αυξήσει περισσότερο την παρουσία της στην Κεντρική Ασία. Προφανώς δεν ξεκίνησε η εμπλοκή μας με την περιοχή αυτή το 2007, αλλά η νέα αυτή στρατηγική έχει δώσει μια σημαντική όψη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο παρούσα στην περιοχή αυτή από ό,τι στο παρελθόν. Κάναμε ένα απολογισμό πέρσι στην ε, κοινή ε, αξιολόγηση Συμφουλίου και κομισιών πέρσι, αυτό ήταν ένα δημόσιο έγγραφο. Θέλω να υπογραμμίσω όμω και μερικά στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν το έγγραφό σα. Όπω ξέρετε, καταρχήν έχουμε υψηλό επίπεδο πολιτικό διάλογο σε τακτικό επίπεδο, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών με τι χώρε τη Κεντρική Ασία, που επέτρεψε σε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζει και πιο ευαίσθητα θέματα, όπω τα θέματα διαχείριση διατήρων πόρων που είναι ιδιαίτερα επίμαχα στην περιοχή αυτή. Επίση, έχουμε διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τι πέντε χώρε τη περιοχή, κάτι το οποίο δεν ήταν εύκολο. Και πρέπει να τονίσουμε ότι κανένα άλλο διεθνή παίκτη στην περιοχή δεν έχει τόσο μεγάλη παρουσία για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο διάλογο αυτό μα έχει επιτρέψει να έχουμε μια συζήτηση σε βάθο επίπεδο εμπειρογνωμόνων και μα επέτρεψε επίση να βρούμε τομεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μεταλαμβαδεύσει την εμπειρογνωμοσύνη τη για να βοηθήσει τι χώρε αυτέ στη διαδικασία μεταρρύθμιση. Φυσικά, εμεί τονίζουμε πάντα σε όλε τι συναντήσει υψηλού επίπεδου τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό συμπεριλαμβάνει και το είπα το επίπεδο όταν γίνονται συναντήσει με του προέδρου των χωρών αυτών. Επίση, στον ενεργειακό τομέα, εμεί τονίζουμε τη σημασία να υπάρξει συμμετοχή στο, για να υπάρξει ένα διάβλος προς την Κασπία και να συμμετάσχει και ο, το Τουρκμενιστάν στον νότιο διάδρομο. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, είχαμε τη δυνατότητα στις συναντήσεις υψηλού επίπεδου να συζητήσουμε <clears throat> ενδελεχώς με τις χώρες αυτές και όλες οι χώρες στον τομέα των υδατινών πόρων προχωρούν τώρα σε ένα διάλογο για τα θέματα αυτά. Και εμείς φυσικά θα συμβάλλουμε όπως έχουμε κάνει και στην Ανατολική Ευρώπη και τον Κάφκασο την εμπειρογνωμοσύνη μας για να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και θα υπάρξει και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη που θα δοθεί από εμά στη μέσω της εκτελεστικής εκτροπή για το Διεθνέ Ταμείο Διάσωση τη Θάλασσα τη Αράλη, που είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο για συνεργασία. Για τα θέματα παιδεία, όπω ανέφεραν και άλλοι ομιλητέ προηγουμένω, όλο και περισσότεροι φοιτητέ έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με προγράμματα ανταλλαγή και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει απόλυτα στην ε, διαδικασία μεταρρύθμιση εκπαίδευση σε ορισμένε χώρε. Σε ό,τι αφορά τώρα την αντιμετώπιση <clears throat> προβλημάτων λαθρεμπορίου και διαχείρισης των ε, συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στα προγράμματα αυτά για καλύτερη διαχείριση των συνόρων και αντιμετώπιση των λαθρεμπόριων και χρειάζεται και περισσότερη διεθνή συνεργασία. Όπω ξέρετε, έχουμε πει στη Ευρύνη την εντολή τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να καλύψει και την Κεντρική Ασία ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη έμφαση στο περιβάλλον και την ενέργεια και έχουμε δημιουργήσει και μια νέα διευκόλυνση επενδύσεων για να υπάρξει και πολλαπλασιασμό τη προσπάθεια Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τονίστηκε και το θέμα των ευρωπαϊκών αντιπροσωπείων στην περιοχή αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε στο Κύρκισταν και το Τατζικιστάν τα τελευταία χρόνια. Θα ανοίξουμε και στην Τασκένδη, στο Ουσμπεκιστάν. <clears throat> για λόγου βέβαια του προπολογισμού υπήρξαν καθυστερήσει <clears throat> για την έναρξη παρουσίαση αντιπροσωπεία στο Τουρκμενιστάν. Ελπίζουμε θα μπορέσει αυτό να γίνει πραγματικότητα σε ένα προσεχές μέλλον. Η κρίση στο Κυργιστάν πέρσι έδειξε την μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από τον Απρίλιο του 2010 που ξέσπασε αυτή η κρίση. Ο κ. Μορέλο, ο δικός μας εκπρόσωπος, ήταν επιτόπου και ξεκίνησε μια διαδικασία συνεργασίας μεταξύ του, της ε, ΟΑΣΕ, του, των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο Κυργιστάν. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία σταθερότητα για να υπάρξει κατασκευή στέγασης στο νότιο μέρος της χώρας αυτής, προετοιμασία του δημοψηφίσματος, προετοιμασία κοινοβουλευτικών εκλογών και τώρα των επικειμένων προεδρικών εκλογών. Όλα αυτά μαζί με την σημαντική μας βοήθεια σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα ένδυα στη χώρα αυτή. Μόλον τούτο, το Κυργιστάν και η ευρύτερη περιοχή αντιμετωπίζουν ακόμα σημαντικέ προκλήσει. Πολλά πρέπει να γίνουν σε σχέση με τι χώρε αυτέ. Όπω αναφέρθηκε από ορισμένου ομιλητέ, η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο εξακολουθεί να είναι ανησυχητικό. Πρέπει να δούμε ποιο μπορούμε εμεί να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο την παρουσία μα στην περιοχή αυτή που είναι τόσο σημαντική και να προωθήσουμε τη δράση τη κοινωνία των πολιτών, η οποία θα είναι σε τελική ανάλυση πάρα πολύ σημαντική για να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην περιοχή αυτή. <clears throat> Είμαστε πεπισμένοι ότι όσο περισσότερο συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή αυτή, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσει να προωθήσει τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω τονίστηκε και από ορισμένου άλλου, εμεί αυτή τη στιγμή με τη διαδικασία εγκατάσταση των αντιπροσωπείων στην περιοχή αυτή, κάτι που θα αυξήσει και την ορατότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο έλειπε στο παρελθόν και θα μπορέσει να βοηθήσει να προωθήσουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα με τρόπο πιο αποτελεσματικό. Λόγω των κάπω περιορισμένων οικονομικών πόρων που έχουμε για την περιοχή αυτή για το 2007 2013 ήταν μονάχα 750 εκατομμύρια ευρώ. Ο συντονισμό των προσπαθειών μα με άλλου διεθνεί χορηγού είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να εντατικοποιηθεί περαιτέρω. Το γεγονό ότι έχουμε περιορισμένου πόρου κάνει πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εστιάσουμε καλύτερα την αρρωγή μα σε ένα μικρότερο αριθμό τομέων όπως παραγωγός χάρη η εξάλληψη της ένδυας που είναι ένα σημαντικό θέμα και για τις φτωχότερες χώρες το Κυργιστάν και το Ταζικιστάν εκεί εστιάζεται το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ μορφή αυτή η περιοχή όπως τονίζει και η εκθέση και παρά το γεγονός ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, διαμεθοριακή συνεργασία σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και συνόρων η κάθε χώρα χρειάζεται μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση η οποία βασίζεται στι διαφορετικές ανάγκες και στις διαφορετικές φιλοδοξίες σε σχέση με την σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τους στόχους μεταρρύθμισης. Για την περίπτωση του Καζακστάν ξεκίνησαν πρόσφατα οι συνομιλίες για μια ενισχυμένη συνεργασία, συμφωνία συνεργασίας και εταιρικής σχέσης. Η Κεντρική Ασία φυσικά βέβαια δεν είναι τμήμα της πολιτικής γειτονίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς μπορούμε να αντλήσουμε εμπειρίες από την ανατολική εταιρική σχέση και από την πολιτική γειτονία όταν αντιμετωπίζουμε τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, αλλά οι χώρες της Κεντρικής Ασίας συμμετέχουν σε μερικά περιφερειακά προγράμματα τα οποία αφορούν την πολιτική γειτονία, παραδείγματο χάρη στον τομέα τη μεταφορά ενέργεια, υδάτινων πόρων και περιβάλλοντο, καθώ και παιδεία. Εν τέλει, μια ακόμα σημαντική πτυχή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τη στρατηγική μα, η οποία κατέστη πάρα πολύ σημαντική λόγω λαμβάνοντα υπόψη και του περιορισμένου πόρου μα, είναι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη χάρη, θεμάτων κράτους δικαίου. Η Γαλλία και η Γερμανία εκεί έπαιξαν ένα πρωτοπόρο ρόλο με την υποστήριξη της Κομισιόν. Η επόμενη φάση τώρα θα εφαρμοστεί από ένα κονσόρτσιουμ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται όλο και περισσότερο σε εμπειρογνωμοσύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ορατότητά μα σε αυτή την περιοχή. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρξει μια μεγαλύτερη εμπλοκή <clears throat> των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσο να πτήσονται περισσότερο οι σχέσει μα με τι χώρε τη Κεντρική Ασία. Θέλω λοιπόν να κλείσω λέγοντα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο καθώ προχωρούμε στι σχέσει μα με την Κεντρική Ασία. Εμεί χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τι επισκέψει των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην περιοχή αυτή και τον διακοινοβουλευτικό διάλογο. Και χαιρετίζουμε και πάλι το σχέδιο ψηφίσματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι είναι μια πολύ σημαντική συμβολή στην επικείμενη αναθεώρηση της πολιτικής μας στην περιοχή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φρίδενσεν. Θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Κίλς Νίλσεν για να μας ε, κάνει μια σύνθεση της συζήτησης. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, που συμμετείχαν στη συζήτηση και βοήθησαν να βελτιώσουμε την έκθεση. Ορισμένες διευκρινήσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν διαπιστώνω ότι συμφωνούμε όλοι για, για τα θέματα του κράτους δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή την περιοχή. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο να διαπιστώνουμε ότι όλοι συμφωνούμε για αυτά τα πράγματα. στην έκθεση ίσως θα, πρέπει να το επαναδιατυπώσουμε στην έκθεση, αλλά ο στόχος είναι εμφανής για να ενισχύσουμε τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην Κεντρική Ασία. Πολλοί συνάδελφοι θεωρούν ότι πρέπει να τονίσουμε ορισμένα σημεία με τα οποία φυσικά εγώ συμφωνώ. Θα δούμε πώς θα το διατυπώσουμε. Ο κύριος είπατε για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στην προστασία, στην προάσπιση των συμφερόντων μας, φυσικά και συμφωνώ μαζί σας. Τώρα για τα σημεία της κυρίας Βέιντερε που ήταν σημεία της κυρίας να δούμε ε, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό χωρίς να προσθέσουμε νέες παραγράφους. Θα το συζητήσουμε, αλλά εγώ φοβάμαι να επανέλθουμε στις 7 προτεραιότητες, γιατί ξαφνικά μπορούμε να αρχίσουμε να προσθέτουμε και αυτό χωρίς να εμπαθύνουμε. Είναι σημαντικό να επιμείνουμε στην προτεραιότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το σεβασμό του δικαίου. Όλοι συμφωνούμε με, αυτό το οποίο, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην, ε, στον αραβικό κόσμο. Ε, πρέπει να τα παλέψουμε αυτά και να τα υποστηρίξουμε. Τώρα, για τον εκπρόσωπο της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων είπε πολλές φορές ότι η Κεντρική Ασία δεν ανήκει στην πολιτική γυτνίαση, αλλά αυτό αιτιολογεί στο να αναλάβει άλλου είδους πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή, διότι πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αρχές μας, ποιες είναι οι προτεραιότητές μας για τα θέματα του σεβασμού του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εντάξει, δεν βρίσκεται στα πλαίσια της πολιτικής γυτνίασης, αλλά πρέπει να δούμε με τη στρατηγική μας τι κάνουμε, ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιος μίλησε, ε, το έχουμε και στην έκθεση, ότι θα πρέπει να βγούμε από αυτήν την στρατηγική που θέλει την σταθεροποίηση των εγκατεστημένων καθεστώτων στην περιοχή, όποια και να είναι η πολιτική τους κλπ. Εγώ απαντώ σε συγκεκριμένες σαφείς ερωτήσεις, εγώ έλαβα υπόψη μου τις προτάσεις και των ΜΕΝ και των ΒΕ, αλλά ο κύριος Πίτερ λέει ε, μου έθεσε μία ερώτηση για το κοινοβουλευτικό φόρουμ. Μα, υποβάλλω μία πρόταση. Εγώ πηγαίνοντας στην περιοχή ε, άκουσα μη κυβερνητικές οργανώσεις να αναφέρουν αυτό το πρόβλημα έλλειψης διαλόγου και ανταλλαγών. Ε, δεν ήταν φυσικά οι αρχές που μου το ανέφεραν. Ε, και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλία με αυτό το κοινοβουλευτικό φόρουμ στην Κεντρική Ασία. Δεν πρόκειται δηλαδή για μία πρόταση των ε, ε, κοινοβουλίων των χωρών αυτών. Μετά βέβαια θα επανέλθουμε σε μια άλλη φάση. Ευχαριστώ κυρία Κύρ Να θυμίσω το χρονοδιάγραμμα κατάθεση για τις τροπολογίες 6 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Η συζήτηση για αυτές τις τροπολογίες θα γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου. 4-5 ε, Οκτωβρίου στην Επιτροπή και στην, τον Οκτώβριο στη δεύτερη Ολομέλεια θα ψηφίσουμε. Πάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης αφορά στη γνωμοδότηση που θα πρέπει να ε, τη γνωμοδότηση προς την Ίντα σχετικά με το πρωτόκολλο συνεργασίας ε, με το Ουζουμπεκιστάν. Αφορά στην επέκταση των διατάξεων της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλώστου υφαντουργικών. Και αυτή η έκθεση για μια χώρα της Κεντρικής Ασίας έχει ως εισηγήτρια την κυρία Κιλ Νίλσεν και εδώ πρόκειται για μια διόρθωση τυπική, αλλά το θέμα του βάμπακος που είναι και η βασική, η βασική είναι που εξάγεται από τη χώρα αποτελεί αντικείμενο ανησυχίας και συνθήκες με τις οποίες παράγεται. Είχαμε μια ιδιαίτερη διαδικασία στην προκειμένη περίπτωση. Είχαμε ένα ψήφισμα για το άρθρο 110 του κανονισμού και δεν επέτρεπε στην Επιτροπή μας να παρέμβει επίσημα σε αυτό το ψήφισμα. Αλλά η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου αποφάσισε σήμερα το πρωί να ε, να συντάξει μια διάμεση έκθεση βάσει του άρθρου 81 του κανονισμού και αυτό μας επιτρέπει να γνωμοδοτήσουμε νομότυπα Οπότε η γνωμοδότηση θα πρέπει να προσαρμοστεί με τη νέα διαδικασία και σχετική ενημέρωση θα σας έρθει με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Θα σας, θα σας αναφέρω το χρονοδιάγραμμα στο τέλος βέβαια. Κυρία Κιλνίλσεν, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, η Καταναγκαστική εργασία των παιδιών είναι μια πρακτική που συνηθίζεται στο Ουζουμπεκιστάν. Είναι μια χώρα δε που είναι και ο δεύτερος εξαγωγέας βάμβακος. Δύο εκατομμύρια μαθητές υποχρεούνται να εργάζονται τρεις μήνες κάθε χρόνο στις βαμβακοφυτίες και αυτό με πολύ δύσκολες συνθήκες το Ουζουμπεκιστάν έχει επικυρώσει τις δύο συμφωνίες της εδώ για την ε, παιδική εργασία, αλλά δεν τη στηρεί. Απορρίπτει συνεχώς το Ουζουμπεκιστάν τις ε, ε, τριμερείς αντιπροσωπείες παρατηρητών της ΔΟΕ και αρνείται συνεχώς τις κατηγορίες που, ε, του ΟΙΕ για την εργασία των ανηλίκων. Εμείς θέλουμε να επιμείνουμε σε αυτόν τον όρο γιατί όταν θα πρέπει να επεκτεθεί η συμφωνία για, τις διμερείς, ε, για το διμερές εμπόριο. Στη Γενέβη η ΔΟΕ ξανακάλεσε την ε, Τασκένδη να δεχθεί κατά την επόμενη σοβιά ε, βαμβακιού ε, την αντιπροσωπεία παρατηρητών αρνήθηκε το Ουζουμπεκίσταν οι μαθητές ε, γυμνασιόπεδα εργάστηκαν το Μάιο στην βασική καλλιέργεια της χώρας 40-45 μέρες σε μια περίοδο πολύ δύσκολη το Μάιο και μάλιστα δύσκολη φάση ανάπτυξης διότι χρησιμοποιούνται ισχυρά χημικά για την καλλιέργεια του Μαμπακιού και θα επανέλθουν τον Οκτώβριο. Η εξαίρεση δε είναι, ανέρχεται στα 60 με 85 δολάρια. Όταν ξέρουμε ότι το κατακεφαλήν εισόδημα στη χώρα είναι 100 δολάρια. Πρόκειται για μεγάλη υποκρισία. Λένε εμείς ε, δεν είμαστε υπέρ της εργασίας των παιδιών, την καταπολεμούμε, αλλά θέτει ποσοστώσει σε κάθε περιφέρεια. Οι κυβερνήτες έχουν μεγάλα βάρη στην πλάτη τους, γιατί είναι υπεύθυνοι για το, ε, για το αποτέλεσμα της ε, <coughs> σοδιάς και υποχρεώνουν λοιπόν τα παιδιά, τους φοιτητές και τους υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους να πηγαίνουν να εργάζονται στους βαβακοφοιτίες. Εμείς θα πρέπει να το απορρίψουμε απόλυτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το σύστημα και την συμφωνία με το Ουζουμπεκιστάν διότι παραβιάζονται ε, εμφανέστατα όλες οι αρχές της ΔΟΕ. Ευχαριστώ κυρία Κιλ Νίλσεν. Η κυρία Βέιτερ έχει το λόγο εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κιλ Νίλσεν για την γνωμοδότησή της, το σχέδιο γνωμοδότησή της, όπως ακούσατε ήδη, έχει δώσει μεγάλη έμφαση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην γνωμοδότηση αυτή και τονίζει την στεναρή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλίσει την αναστολή του διμερούς εμπορίου κλωστοεφαντουργικών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουσμπεκιστάν μέχρι ότου ανεξάρτητοι διεθνείς εμπειρογνώμονες διαπιστώσουν την κατάσταση για τους εργαζόμενους στα κλωστοεφαντουργικά στη χώρα αυτή. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι η δημοκρατία του Ουσβεκιστάν είναι εταίρος μας. Έχουμε, έχουμε συνάψει μια συμφωνία με τη χώρα αυτή, η οποία έχει συνεργαστεί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλά προγράμματα ανάπτυξης ε, στον τομέα αυτό. Το να αναστείλουμε τη συνεργασία αυτή θα σήμαινε ότι θα κάνουμε κατάχρηση ενός από τα πιο σημαντικά μας εργαλεία της ε, συνεργασία στον οικονομικό και εμπορικό τομέα. Η οικονομική και η κοινωνική ανάπτυξη και η δημοκρατία είναι αλληλένδετες. Έχουμε πολύ περισσότερε δυνατότητε να προωθήσουμε την ανάπτυξη και τη δημοκρατικοποίηση στο Ουσμπεκιστάν και να ενισχύσουμε τη διμερή συνεργασία σε άλλα θέματα διατηρώντα αυτή τη συνεργασία, όπω είναι παραδείγματο χάρη τα θέματα ασφάλεια τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ουσμπεκιστάν. Αυτά όμως υπό την προϋπόθεση ότι θα είμαστε ένα εταίρος ο οποίο θα τηρήσει τα υπεσχημένα και όχι να τα ε, παραγνωρίσει. Επίσης, η διακοπή της συνεργασίας θα δημιουργήσει οικονομικά προβλήματα στον πληθυσμό του Ουσμπεκιστάν που εξαρτάται τα μάλα από την παραγωγή του βάμβακος. Επίσης, όπως ξέρουμε και από την προσωπική μας ε, εμπειρία και από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, η ρητορική δεν έχει τύχει μεγάλης και θετικής αποδοχής από το Ουσβεκιστάν. Δεν πρέπει λοιπόν να κάνουμε τους γυμνασιάρχες αν θέλουμε να επιτύχουμε κάτι στην περιοχή αυτή. ιδίω όταν υπάρχει η παρουσία μεγάλων δυνάμεων όπως η Ρωσία και η Κίνα, εμείς θα πρέπει να έχουμε μια πιο φιλική στάση προς το Ουσβεκιστάν. Θα πρέπει να αποφύγουμε επίσης και τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Βλέπουμε πόσο μεγάλε είναι οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία που δεν θεωρούνται θετικές συνθήκες, αλλά κανείς δεν θεωρεί ότι πρέπει να αναστείλουμε το εμπόριό μας με τη Ρωσία. Επομένως, δεν θα πρέπει εμείς να εγκαταλείψουμε τους εταίρους μας χωρίς να, να αναγνωρίσουμε αυτά τα οποία έχουν επιτύχει μέχρι στιγμής. Το Σμπεκστάν έχει κάνει πρόοδο βαθμία για να υπάρξει μια νομοθεσία η οποία απαγορεύει την καταναγκαστική και παιδική εργασία εν κατακλείδη. Νομίζω ότι πρέπει να εγκρίνουμε το πρωτόκολλο αυτό, το οποίο θα παρατείνει την διμερή συνεργασία με το Ουσμπεκιστάν εφόσον περιλαμβάνει και ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας κατά της καταναγκαστικής εργασίας ή πρακτικών που θέτουν την ε, υγεία και την πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών εν Μια συνεχιζόμενη παρακολούθηση από την ΔΟΕ και την UNICEF των συνθήκων στο Ουσβεκιστάν είναι απαραίτητες για να μπορούμε να έχουμε μια πλήρη παρακολούθηση της επιτόπιας κατάστασης. Αυτή είναι λοιπόν η απόψή μου και σας ευχαριστώ που με ακούτε. Σας ευχαριστώ ο κύριος είναι για την σοσιαλιστική ομάδα. Ευχαριστώ εκ μέρου τη Μαριλένη Κοπά που πρέπει να, έπρεπε να είναι σε μια άλλη συνεδρίαση. Μιλάω εδώ σήμερα. Είναι ένα δύσκολο θέμα και δεν θα είναι εύκολο να πάρουμε κάποια απόφαση. Όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις οδηγίες που θα δώσουμε εμείς ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Δεν μπορούμε απλώ να δώσουμε ένα πράσινο φως για να υπογραφεί το πρωτόκολλο αυτό. Είναι σημαντικό να μην δείχνουμε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στις σχέσεις μας με τρίτες χώρες. Επίσης, η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουσμπεκιστάν, ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα με την καταναγκαστική παιδική εργασία, είναι κάτι που πρέπει να μας οδηγήσει να συνεχίζουμε το διάλογο με τις αρχές εκεί. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να επιμείνουμε το Ουσμπεκιστάν να επιτρέψει στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ελεύθερα να μπορέσει να επισκεφθεί τη χώρα, να ελέγξει και να δει πώς έχει η κατάσταση εκεί όσον αφορά την κατανακαστική εργασία η θέση της κυβέρνησης του Ουσβεκιστάν μέχρι τώρα ήταν να αρνείται το πρόβλημα. Οι πληροφορίες όμως που εμείς έχουμε είναι ότι υπάρχει το πρόβλημα, παραμένει. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει απαγόρευση καταναγκαστικής εργασίας στην νομοθεσία του Ουσβεκιστάν. Έτσι λοιπόν το θέμα αυτό πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να ελεγχθεί εκ νέου πριν δοθεί το πράσινο φως για να υπογράψουμε το πρωτόκολλο. Ένα άλλο θέμα που πιστεύω ότι είναι σημαντικό βάσει εκθέσεων που μας έρχονται από μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι η χρήση ύδατος στις βαβακοκαλλιέργειες, ότι δηλαδή χρησιμοποιούνται οι φυσικοί πόροι με τρόπο μη ορθολογικό. Είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε με τις αρχές. Η Επιτροπή, ίσως και το Συμβούλιο θα μπορούσαν να αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες. Αυτή είναι η θέση της ομάδας μας όσον αφορά τη χρήση δάτων. Ευχαριστούμε κύριο Μπρόκ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας συγχαρώ για την, ε, το σχέδιο γνωμοδότησή σας. Εγώ δεν ήξερα ο ίδιος πόσο μεγάλη είναι η έκταση της παιδικής εργασίας που τονίζετε στην έκθεσή σας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να μας δώσετε και την έκθεση της Διεθνής ε, Οργάνωσης Εργασίας. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον να γνωρίσουμε τι ακριβώς αναφέρεται στα θέματα αυτά. Όταν διαπραγματευόμαστε με αυτά τα κράτη και όταν εμπλέκονται και εμπορικά θέματα θα πρέπει να γνωρίζουμε αν υπάρχουν πραγματικά παραβιάσεις των διεθνών προτύπων για την εργασία του, της ΔΟΕ κτλ. Ίσως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και στο διευρυμένο, στη, στη συνάντηση του διευρυμένου Προεδρείου. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη <clears throat> εφαρμογή των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι τη χρήση δύο μέτρων και δύο σταθμών. Να υπάρξει λοιπόν καλύτερη συνεργασία με την ε, Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου και να έχουμε επομένως μια πιο αποτελεσματική ε, εφαρμογή των αρχών μας σε επίπεδα διεθνής πολιτικής, εκεί ιδίω που έχουμε περιορισμένες δυνατότητες δράσης. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να εξασφαλίσουμε το κατά πόσο μπορούμε να διαπιστώσουμε και ποιε επιχειρήσει οι οποίε προερχόνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζοντα την κατάσταση τη παιδική εργασία στο Ουσμπεκιστάν, παρόλα αυτά ε, χρησιμοποιούν τον παραγόμενο βάμβακα στο Ουσμπεκιστάν. Αυτό είναι ενδιαφέρον να το γνωρίζει και ο καταναλωτής φυσικά αυτού του βάμβακος για να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση στις επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν το βάβακα από το Ουσπεκιστάν. Αυτά μπορούν να αυξήσουν λοιπόν και την πίεση η οποία μπορεί να ασκηθεί και να ευνοήσουν μια <clears throat> καλύτερη συνειδητοποίηση και μεγαλύτερη εφαρμογή της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ε, εμπορικές μας συμφωνίες. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να θέσουμε και το θέμα μια κοινή έκθεση με την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου για να εξασφαλίσουμε την κοινή εφαρμογή των προτύπων μα σε τέτοιε διεθνεί συμφωνίε. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπρόκ. Πρώτα απ' όλα θα, σας, ε, θα διανύμουμε σε όλους αυτή την έκθεση της, του, της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας <clears throat> και επίσης το Σεπτέμβριο θα είναι παρόντε και οι εκπρόσωποι τη UNICEF στο Ουσβεκιστάν. Θα οργανώσουμε μια συνάντηση με αυτού και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι απόψει του και να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί του. Και για να απαντήσω σε αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριο Μπροκ, η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου ασχολείται και αυτή με τα πρότυπα ε, σε ό,τι αφορά την εργασία. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια, θα ήταν πολύ υποφελής μια ανταλλαγή, μια συνεργασία μαζί τους και ιδίως για τα θέματα παιδικής εργασίας όπου έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες. Την τώρα το λόγο στον κύριο Σβόμποντα, ο οποίο ζήτησε το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θέλω να υποστηρίξω απλώς αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπροκ. Γιατί πολλοί από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η παιδική εργασία και θέλουν να μην υπάρχει υποστήριξη από τις επιχειρήσεις αυτής της ε, δραστηριότητας τονίστηκε στο Ουσμπεκιστάν ότι υπάρχει μια δυσκολία να υπάρξει ο έλεγχος αυτής της εργασίας γιατί πολλές φορές γίνεται από τις οικογένειες. Ε, αλλά όταν αυτό γίνεται σε μια φάση που τα σχολεία λειτουργούν, εκεί πέρα αυτή πρέπει να είναι μια τελείως αξιόπινη δραστηριότητα. Είναι απαραίτητο, όπως είπατε, να προσκαλέσουμε τους εκπροσώπους της ΔΟΕ και της ε, UNICEF και αυτό μπορεί να είναι η, η ευκαιρία να το πράξουμε στην περίπτωση του Ουσμπεκιστάν, αλλά θα πρέπει να θέσουμε και ένα γενικότερο θέμα. Εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παιδική εργασία να γίνουν σεβαστά σε διεθνές επίπεδο και να τονίζεται η σημασία τους σε όλες τις ε, συμφωνίες που, συν, ε, που στις οποίες εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό επομένως θα είναι μια πρωτοβουλία την οποία μπορούμε να υποστηρίξουμε. Δίνω και πάλι το λόγο στον κύριο ένα από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να αναφερθώ λίγο στην παιδική εργασία. Ίσως και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή να έχουν κάτι να πούν. Συζητήσαμε και νωρίτερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όντω αποτελούν κεντρικό σημείο στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και γενικότερα. Σε διάφορες συζητήσεις που έχουμε σε ανώτατο επίπεδο το συζητάμε. Συζητάμε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά. Και είναι θέματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με το Ουσπικιστάν, αλλά σίγουρα και με το Ουσπικιστάν. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες ε, που εκφράζονται στις επαναλαμβανόμενες εκθέσεις του Διεθνούς, ε, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όσον αφορά την ε, παιδική εργασία και στη συνεδρίασή μας τον Ιούλιο στο, εδώ στις Βρυξέλλες που είχαμε με ομολόγους μας το συζητήσαμε και το θέσαμε. Η UNICEF είναι καλή να προσκληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η UNICEF έχει πρόσβαση και μπορεί να ελέγξει το τι γίνεται στις καλλιέργειες βαμβακιού. Οπότε είναι καλό να μιλήσουμε μαζί τους. Όπως είπανε και κάποιοι, κάποια θετικά βήματα έχουν γίνει στο Σβεκιστάν. για παράδειγμα η νομοθεσία ε, της χώρας, η οποία απαγορεύει την ε, παιδική εργασία και προσπαθεί να συμμορφωθεί με ε, τις διατάξεις και τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Όντω λοιπόν γίνονται προσπάθειες, παρόλα αυτά υπάρχει καταναγκαστική εργασία. Πρέπει να πιέσουμε για να εφαρμοστεί και στην πράξη βέβαια η νομοθεσία της χώρας. Τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί κάπως ο αριθμός των παιδιών. Βέβαια εμείς θέλουμε να δούμε ακόμα περισσότερα. Μην παραβλέπουμε όμως και τα κάποια θετικά και σίγουρα να πιέσουμε το Ουσπεκιστάν να δεχθεί την επίσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στις βαμβακοκαλλιέργειες για να ελέγξει ε, τα πράγματα επιτόπου. Σίγουρα χρειάζεται και ο πολιτικός διάλογος ε, και βοήθεια γενικότερα, αλλά να πιέζουμε για βελτίωση της κατάστασης. Τεχνική αρρωγή επικεντρώνεται στην βελτίωση του επίπεδου ζωής στην Ήπεθρο της χώρας. Αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε και σίγουρα πρέπει να βοηθήσουμε και για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες εκπαίδευση κλπ. Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη της υπαίθρου είναι κάτι που σίγουρα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και να βοηθήσει και στο θέμα της παιδικής εργασίας. Νομίζουμε λοιπόν ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι να συνεχίσουμε να ζητάμε και να πιέζουμε τις αρχές του Ουσπεκιστάν για να λυθεί το πρόβλημα της παιδικής εργασίας. Με συνεργασία ε, με την ε, Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Θα επιμένουμε πάνω σε αυτό. Είπαμε, έχουν γίνει ήδη κάποια βήματα στο Ουσπεκιστάν, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας μαζί τους, γιατί μια τέτοια προσέγγιση συνεργασία είναι ο καλύτερο τρόπο για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. Η κυρία Κιλνίλσεν ε, τώρα, η συγγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ενημερώσω του συναδέλφους ότι είχα την ευκαιρία πολλές φορές μέχρι τώρα να πάω στην Επιτροπή. Τα πήρα και το λόγο, ανταλλάξα απόψει μαζί τους. Και διευκρινίζω ότι επί του παρόντος ε, δεν, ότι πρέπει να, δεν λένε ότι πρέπει να αρνηθούν την συμφωνία αυτή, αλλά η Επιτροπή Ίντα ζητάει τα αποτελέσματα της αποστολής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας να δημοσιευθούν και μετά από αυτό θα αποφανθούν. Γι' αυτό λοιπόν εμείς επιμένουμε να υπάρξει αποστολή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στο Ουσβεκιστάν και περιμένουμε τα αποτελέσματα από μια τέτοια αποστολή. Αυτό που πιστεύω ότι είναι σημαντικό είναι για τη UNICEF. Πράγματι συναντήθηκα με εκπροσώπους της UNICEF στο Ουσβεκιστάν και ξέρω τι δουλειά κάνουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή είναι μια δουλειά που όντω επέτρεψε να μειωθεί η παιδική εργασία εκεί. Βελτιώθηκε η αποτελεσματικότητα, δηλαδή η απόδοση των ε, ενηλίκων που εργάζονται στις βαβακοκαλλιέργειες. Όντω είναι καλό να συναντηθούμε με τη UNICEF. Και προτείνω, αν συμφωνείτε, το εξή. Μια μήνυα ακρόαση με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την ίντα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε όλοι μαζί κάτι για την παιδική εργασία. Θα ήταν ενδιαφέρον και θα μας επέτρεπε να προχωρήσουμε κάπως. Όντως υπάρχει κάποια πρόοδος σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Το γνωρίζω, ξέρω ότι δουλειά γίνεται εκεί από τη UNICEF. Αλλά γι' αυτό δεν πρέπει να σταματήσουμε να συνεχίζουμε την πίεσή μας. Και πρέπει να επιμείνουμε ώστε τα πράγματα να πάνε ακόμα πιο μακριά. Πρέπει να επιμείνουμε επίσης για... στο εξή, στο ότι η κυβέρνηση έχει την υπευθυνότητα. Δεν μπορεί να βάζει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορεί από τη μια να λέει, μα κοιτάξτε εμεί έχουμε απαγορεύσει την παιδική εργασία και από την άλλη μεριά, εγώ όντω χρησιμοποιώ τον όρο υποκρισία, από την άλλη μεριά υποκριτικά να επιμένει ε, για μεγαλύτερη απόδοση ε, στη σοδιά. Αν λοιπόν ε, συμφωνείτε κι εσείς, Ας οργανώσουμε αυτή την κοινή ε, μήνυα ακρόαση την οποία σας ανέφερα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κιλ Νίλσεν. Υπενθυμίζω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τώρα. Ε, δεδομένων των προθεσμών που έχουμε για την έγκριση της έκθεσης και πότε θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια, προτείνω το εξή. Και παρακαλώ τις τροπολογίες σας, τα αγγλικά μόνο παρακαλώ. 6 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών θα συζητήσουμε στις 12 ε, Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο και η Ίντα μετά θα ψηφίσει και στη δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου, λέει η Πρόεδρος, θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Τώρα, περνάμε στην ε, θέση της ε, Επιτροπής μας όσον αφορά την ε, τελική έκθεση της Επιτροπής Προπολογισμών για τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού του 2012. 12 ε, Σεπτεμβρίου θα τροποποιήσουμε την ε, έκθεση αυτή και έτσι θα καταλήξουμε στη θέση ΑΦΕΤ που ελπίζουμε να αντικατοπτριστεί στην έκθεση της Επιτροπής Προπολογισμών. Εισηγήτρια για 10 λεπτά και μετά οι σκιώδες εισηγήτες θα πάρουν το λόγο. Κυρία Μούνη, θα έχετε το λόγο. Δεν με ακούει όμως η κυρία Μουνίθ. Παρακαλώ, κύριε Μουνίθ, έχετε το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που δεν σας άκουγα. Έρχομαι λοιπόν στο σημείο αυτό του προϋπολογισμού. Θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές και όλους αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν με τροπολογίες και άλλες επικοδομητικές συνεισφορές για, την, ε, για τις τροπολογίες και την ε, λίστα ψηφοφορίας, <clears throat> ώστε να έχουμε μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία να είναι συμβατή και συνεκτική και με τις πολιτικές μας προτεραιότητες που ενεκρίθησαν το Μάιο και με την κατάσταση περιστολής των πόρων που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Να σας δώσω μονάχα ένα αριθμητικό στοιχείο. Ο προϋπολογισμός έχει μειωθεί κατά 2,2% 350 εκατομμύρια σε πιστώσεις πληρωμών και 90 εκατομμύρια σε πιστώσεις υποχρεώσεων είναι η μείωση του προπολογισμού που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για τα θέματα εξωτερική δράση. Λοιπόν, έχουμε μια κατάσταση λιτότητα και περιορισμών που σημαίνει 103 εκατομμύρια σε επιστώσει πληρωμών και 90 σε πιστώσει υποχρεώσεων σε σχέση με την αρχική πρόταση τη Κομισιόν. Επομένω, 2% η μείωση των πιστώσεων πληρωμών και 5,5% δύο Αύξηση της πιστώσης υποχρεώσεων. Αυτό ανταποκρίνεται δεν ανταποκρίνεται μάλλον στην αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρχουν νέες ε, πιστώσεις για να αντιμετωπίσουμε τις νέες υποχρεώσεις που έχει να αντιμετωπίσει το, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε παραγωγικά τις πολιτικές που έχουν να κάνουν με τη Μεσόγειο, τις πολιτικές που έχει θεσπίσει η Επιτροπή μας ήδη το Μάιο. Είναι σαφές λοιπόν ότι θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία των υποχρεώσεων αυτών και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι ο εκτελεστής των πολιτικών αυτών, θα πρέπει να κατανοήσει καλύτερα και ποιες είναι οι, οι απαιτήσει της υλοποίησης αυτών των πολιτικών σε επίπεδο προϋπολογισμού και εμείς επομένως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τη σημασία των προγραμμάτων που έχουν πολιετή χαρακτήρα, όπου είναι απαραίτητο η Κομισιό να μας πει ποια είναι οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν, ποια είναι η εμπειρία απορρόφησης σε πολιετές επίπεδο. Έχουμε λοιπόν νέε ανάγκε δαπανών, έχουμε μείωση των πόρων, η ανάγκη να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τι πολιτικέ μα προτεραιότητε και έχουμε φυσικά και τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει εκφραστεί μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη προτεραιότητα στα κονδύλια τα οποία αφορούν την πολιτική για την νότια οχθή της Μεσογείου, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της δικής μας Επιτροπής θα τεθούν ένα αμφιβόλο αν δεν μπορέσουμε να σεβαστούμε τις υποχρεώσεις που έχουμε ε, αναλάβει στο παρελθόν. Δεν μπορούμε λοιπόν να λαμβάνουμε νέες προτεραιότητες και να παραγνωρίσουμε τις προηγούμενες προτεραιότητες με τον τρόπο αυτό. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτή την αρχή σε σχέση με την αντιμετώπιση των περιορισμών κονδυλίων που ζητά το Συμβούλιο. Εμεί έχουμε θεσπίσει μια σειρά από κριτήρια, τα οποία νομίζω ότι μπορούν να γίνουν αποδεκτά από όλα τα μέλη τη Επιτροπή μα, γιατί πρόκειται για στόχου οι οποίοι είναι εκείνοι και αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εκπόνηση του καταλόγου ψηφοφορία και των τροπολογιών. Η Κομισιόν φυσικά είναι αυτή η οποία είναι αρμόδια να αξιολογήσει τις συγκεκριμένες ανάγκες για κονδύλια σε περιοχές που δεν περιλαμβάνει δεν περιλαμβάνονται στην ε, δική μας, στις δικές μας προτεραιότητες, αλλά θα πρέπει να αξιολογήσουμε και εμείς σωστά τις προτεραιότητες αυτές και γι' αυτό επανερχόμαστε στο σχέδιο που προπολογισμού για τις γραμμές αυτές. Κατά δεύτερο, οι γραμμές που αφορούν σε προτεραιότητες της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων είναι εξής θα πρέπει να αποκαταστήσουμε τα ποσά του 2011 στην περίπτωση που αυτά τα ποσά είναι υψηλότερα από την πρόταση της Κομισιόν στο σχέδιο προϋπολογισμού και που μειώθηκαν από το Συμβούλιο για να χρηματοδοτήσει νέες προτεραιότητες με αυτά τα κονδύλια, δηλαδή τη Μεσόγειο. Εμείς πρέπει να είμαστε σαφείς σε αυτό το τομέα και να υποστηρίξουμε το υψηλότερο δυνατό ποσό, αυτά του 2011 σε περίπτωση δηλαδή που αυτά τα ποσά είναι ψηλότερα από την πρόταση της Κομισιόν. Ένα άλλο κριτήριο που είναι θεμελιώδες και θα σας εξηγήσω τώρα και το σαφές περιεχόμενο του καταλόγου ψηφοφορίας και των ε, τροπολογιών. Εμείς στον προπολογισμό θα πρέπει να αντικατοπτρίζουμε τις θέσεις του Κοινοβουλίου έτσι όπως πέρασαν από ψηφίσματα και, από, και τις θέσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Αναφέρομαι εδώ στην, στο άνοιγμα των γραφείων των αντιπροσωπιών των εξωτερικών, ε, της εξωτερικής ε, δράσης κλπ ο συνάδελφος Γκουαλτιέρη ασχολήθηκαν και άλλοι συνάδελφοι από άλλες ομάδες ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα πιο συγκεκριμένα αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να επισημάνουμε ποιο είναι το φύλλο πορείας για την εγκατάσταση και την επέκταση των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε μία αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο των Χωρών του Κόλπου και στο Ιράν. Το ζητάμε αυτό με ψηφίσματα του Μαρτίου του 2011. Εμείς αυτά τα ποσά τα έχουμε βάλει στο αποθεματικό ούτω ώστε να υπάρχει ένα κάποιο κίνητρο προς την Κομισιόν για να αρχίσει να ετοιμάζει τις ε, αντίστοιχες αποφάσεις. Η εφαρμογή αυτών των κριτηρίων προϋποθέτει ότι εγώ είμαι κατά των τροπολογιών εκείνων που μειώνουν τα κονδύλια των γραμμών προτεραιότητας, όπως εκφράζονται από την Επιτροπή μας, που μειώνουν τα ποσά του 2011 στις γραμμές εκείνες που δεν είναι προτεραιότητες αλλά που η Επιτροπή έχει ορίσει ποιες είναι οι ανάγκες της ως προς τις δαπάνες. Τώρα, για τις τροπολογίες που θέλουν να αυξήσουν γραμμές οι οποίες να αυξήσουν υπέρμετρα γραμμές οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα ε, πολιτικό νόημα να χρηματοδοτούν τόσο υπερβολικά και που ε, δεν έχουν και σχέση και με το πρεστίζ του Κοινοβουλίου. Τώρα θέλω πέντε λεπτά για να σας εξηγήσω τη γενική γραμμή και τις τροπολογίες. Πρώτη κατηγορία. Σε εκείνες τις γραμμές στις οποίες εμείς αποκαθιστούμε τα ποσά της Κομισιόν στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε βοήθεια και θεσμική επικουρία στις υποψήφιες χώρες αποκαθιστούμε λοιπόν το ποσό της Κομισιόν που είναι υψηλότερο από εκείνο του 2011 και είμαστε κατά των τροπολογιών ε, μείωσης. Οριζόντια και τα προγράμματα και εδώ είμαστε κατά των θέσεων του Συμβουλίου, δηλαδή τροπολογίες ε, Σαλαφράγκα 50, 18, 50 δεν θα σας ε, κουράσω αναφέροντάς σας ε, ακριβώς ποιος είναι ο αριθμός των τροπολογιών. Τώρα συνεργασία με τις τρίτες ε, βιομηχανημένες χώρες, απάντηση στην κρίση, καταπολέμηση βιολογικών, χημικών, ατομικών κινδύνων. Είναι ένα θέμα το οποίο δημιούργησε εδώ συζήτηση αφορά στο θέμα της ε, βοήθειας ε, ανοικοδόμησης του Αφγανιστάν και χαίρομαι που είναι εδώ ο κύριος Αρλάκη. Εμείς αποκαθιστούμε την πρόταση της Κομισιόν στον προϋπολογισμό 2011. Υπάρχει μία εγκάρσια τροπολογία του κυρίου Αρλάκη και άλλων πολιτικών ομάδων που θέλουν να αυξηθεί κατά 50 εκατομμύρια ευρώ η γραμμή για την αντικατάσταση των καλλιεργών οποίου, οποίου με εναλλακτικέ καλλιέργειες. Επί της ουσίας συμφωνούμε, αλλά στην κατάσταση που είμαστε σήμερα με την ε, δημοσιονομική λιτότητα δεν, έχει, δεν νομίζω ότι θα περάσει ποτέ κάτι τέτοιο από την Επιτροπή Προϋπολογισμών ούτε και η Κομισιόν θα μπορέσει να το διαχειριστεί όλο αυτό στο εφαρμοστικό του πεδίο, δηλαδή άμα περάσει μια τέτοια πρόταση. Εγώ ζητώ λοιπόν να έχουμε μία τροπολογία, να διατηρεί δηλαδή το 2000, τον προπολογισμό του 2011, ανώτερο δηλαδή από την πρόταση του Συμβουλίου. Και να έχουμε και μερικά σχόλια στη γραμμή που να προτείνει αυτή την εγκάρσια τροπολογία, δηλαδή μέρος αυτών των κονδυλίων να ε, το αφιερώσουμε για την αντικατάσταση των καλλιεργών ε, οποίου με άλλες καλλιέργειες. Αντί δηλαδή να ζητήσουμε αυτή την υπερβολική αύξηση, έστω και αν συμφωνούμε επί της ουσίας. Συνεργασία Ιράκ, Ιράν, Ιεμένη. Εμεί πάλι αποκαθιστούμε το σχέδιο προϋπολογισμού της Κομισιόν 3 ε, εκατομμύρια παραπάνω από την πρόταση του Συμβουλίου. Το ίδιο και με τη συνεργασία με την Ασία. Πάλι εδώ έχουμε το σχέδιο προϋπολογισμού που ισχύει το 2011 ήταν ψηλότερο το ποσό, αλλά τότε η συνεργασία με την Ασία δεν ήταν μεταξύ των προτεραιοτήτων της Επιτροπής, όπως εκφράστηκαν το Μάιο άλλο που είναι συμβατό με τις προτεραιότητες είναι η αποστολή παρατηρητών σε εκλογές. Ζητάει να περικόψουμε κατά 3 εκατομμύρια το Συμβούλιο. Η συνεχής ε, υποστήριξη για την εποπτεία εκλογών εκ μέρους του Κοινοβουλίου και το βεβαρημένο ε, χρονοδιάγραμμα που έχουμε, ε, εκλογικό χρονοδιάγραμμα, μας οδηγεί να υποστηρίξουμε την τροπολογία Λάμψφορτ αλλά και τη δική μου για να μπορέσουμε να έχουμε αυτόν τον προπολογισμό, τον αρχικό δηλαδή. Άλλο, Παλαιστίνη. Τόσο το Συμβούλιο όσο και η Κομισιόν πρότειναν να μειώσουμε κατά 100 εκατομμύρια ευρώ έναντι του 2011. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε για την ειρηνευτική διαδικασία, την βοήθεια στους πρόσφυγες και την ενίσχυση στην Παλαιστινιακή Αρχή αυτά τα ποσά. Το ποσό είναι 300 εκατομμύρια ευρώ και τελικά το δεσμευόμενο ποσό είναι 350, 350 ε, εκατομμύρια. Υποστηρίζουμε λοιπόν τις τέσσερις διαφορετικές τροπολογίες που ζητούν να αυξήσουμε αυτά τα κονδύλια. Έχουμε μία εγκάρσια τροπολογία των διαφόρων πολιτικών ομάδων που ζητούν να έχουμε δύο χωριστές γραμμές για την ενίσχυση για την Παλαιστινιακή Αρχή και μια άλλη γραμμή πιο συγκεκριμένη για τη βοήθεια στους πρόσφυγες. Τόσο εγώ όσο και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι θα συναντηθούμε με την Κομισιόν και με την ουρώ για να δούμε πώς θα διαπραγματευτούμε ακριβώς την γραμμή. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ο συντονισμός μεταξύ Ηνωμένων Εθνών, Παλαιστινιακής Αρχής, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της του Οργανισμού για τους Πρόσφυγες είναι πολύ καλή. Δεν χρειάζεται να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο κονδύλια. Και αυτή η τροπολογία που ζητεί να ξεχωρίσουμε, να σπάσουμε τη γραμμή σε δύο, θέλει την έκπτωση του Συμβουλίου των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, εδώ δεν πρόκειται όμως για κάτι το ιδιαίτερα λειτουργικό, ούτε η Ούρα μας το έχει ζητήσει. Εγώ λοιπόν θεωρώ, εφόσον δεν συντρέχει λόγος, ότι θα πρέπει να την απορρίψω αυτήν την τροπολογία. Δεν τη δέχομαι έστω και αν είναι μια εγκάρσια τροπολογία από πολλές πολιτικές ομάδες. Πάντα όμως εμείς μπορούμε να βρούμε φόρμουλες, τρόπους δηλαδή για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τώρα, στην αρχή βέβαια η πρόταση ήταν να μπουν όλα στο αποθεματικό. Διότι θέλαμε να βοηθήσουμε την ειρηνευτική διαδικασία ξεπερνώντας αυτό το πλαίσιο της παροχής βοήθειας και μόνο. Βέβαια αυτό πρόκειται για κάτι το ευκταίο, δεν μπορούμε να το πετύχουμε με τον προϋπολογισμό. Πάντως πραγματικά πρέπει να, βρούμε τρόπους ε, πιο εφάνταστους ε, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αποτελεσματικότερα στην επίλυση του προβλήματος, το οποίο μένει εκεί στατικό. Για το Easy Plus εμείς έχουμε πάλι τα 16 εκατομμύρια του 2011 με την τροπολογία Σαλαφράγκα και τη δική μου συνεργασία με τη Λατινική Αμερική να σας πω μερικά πράγματα. Αυτή η γραμμή πραγματικά περικόπτεται δίπλα. Έχουμε 25 εκατομμύρια ευρώ τα οποία περικόβονται από το 2011 και μετά στο 2011 είχαμε και μία επανατοποθέτηση των κονδυλίων 26 εκατομμύρια δηλαδή. Λοιπόν, κύριε, θα ήθελα ο κύριος Μπρόκ και ο συνομιλητής του να μην φωνασκούν. Οι 26 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν δόθηκαν αλλού και δεν μπορέσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τη γραμμή της Λατινικής Αμερικής, διότι τα πήραν τα λεφτά και τα βάλανε στη Μεσόγειο. Τι σημαίνει αυτά. Τα 367 εκατομμύρια που τα εγκρίναμε στο οικονομικό έτος 2011. Είχαμε εγκρίνει αυτό το ποσό διότι είχαμε θεωρήσει τόσο η Κομισιόν όσο και εμείς ότι ήταν απαραίτητο. Για να καλυφθούν οι ανάγκες της Λατινικής Αμερικής και περικόπηκαν στα 352 με αυτό το διορθωτικό που μας παρουσίασε η Κομισιόν. Και δεν υπάρχει καμία συνέχεια. διότι δεν έχουν αλλάξει τα ζητούμενα που είχε θέσει αυτή η Επιτροπή, ούτε και οι διαπιστώσεις σχετικά με τις προτεραιότητες. Και βασιζόμενοι στο κριτήριό μας και πάντοτε υπό το φως της λιτότητας ζητάμε να αποκατασταθεί το ποσό του 2011 και προσθέτουμε και τα 26 εκατομμύρια τα οποία τα βγάλανε χωρίς να μας διαβουλευθούν. Και αφού δεν μας ρωτήσανε ζητούμε να τα ξαναβάλουν τα 26 εκατομμύρια. και θέλω να σας πω, να σας εξηγήσω τα πράγματα και κάπως ε, και άλλα επιχειρήματα δηλαδή να μην νομίζετε επειδή είμαι Ισπανίδα ότι με καίει η Λατινική Αμερική διότι κάθε φορά που μιλάνε οι Ισπανοί για Λατινική Αμερική είναι σαν να μιλάμε για τάβρους ε, λοιπόν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί μέσα στην ίδια δημοσιονομική γραμμή εμείς δεν αρνούμεθα ότι οι σχέσεις με τη Βενεζουέλα δεν πληρούν τους όρους για την ε, ανάθεση των κονδυλίων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα ποσά τα οποία δεν τα δίνουμε στη Βενεζουέλα πρέπει να τα παίρνουμε να τα δίνουμε αλλού. Θα έπρεπε πρώτα να ψάξουνε να ψάξουν πού θα μπορούσαν να δώσουν τα λεφτά. Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων, ας πούμε, στην Πενεζουέλα, τότε να ψάχνει κανείς αλλού, στην ίδια περιοχή. Και μετά, θα έπρεπε κανείς να ψάξει να δει άμα η όλη ευελιξία έπρεπε να περάσει σε άλλες γραμμές ή όχι. Οποιαδήποτε λοιπόν κίνηση ή τροποποίηση των ποσών που έχουμε με το οποίο έχουμε πρικοδοτήσει τις γραμμές του προϋπολογισμού, δεν θα πρέπει να γίνεται αφερετα Πρέπει να υπάρχει διαβούλευση. Και το λέω δηλαδή για να το ξέρετε, για προειδοποίηση. Όχι επειδή δηλαδή πρόκειται για τη Λατινική Αμερική να νομίζετε ότι με καίει, Και εντάξει, πήραν τα λεφτά και χρηματοδότησαν την Μεσόγειο, αλλά σήμερα κόβουν την ε, Λατινική Αμερική, αύριο θα το βγάλουν από τη Συμφωνία σταθερότητα και πάει λέγοντας και θα αρχίσουν να βγάζουν όπου θέλουν. Τελευταίο και τελειώνω. Παρουσιάσαμε τέσσερις προπαρασκευαστικές δράσεις με σχέδια πιλότο. Η ε, συμφωνία όλων των πολιτικών ομάδων τα έχετε στα έγγραφα. Και υπάρχει μία τροπολογία που ελπίζω να υποστηριχθεί από την ομάδα για τη νέα διάρθρωση για τις ε, γυναίκες στα πλαίσια των, ε, του ΟΗΕ και των διαφόρων περιοχών για την ισότητα των φύλων και επίσης υποστηρίζουμε τις τροπολογίες της κυρίας Γκόμες και άλλων σχετικά με τη βία κατά των παιδιών και των γυναικών. Ευχαριστώ και πάλι τη γραμματεία της Κομισιόν, τους βοηθούς μου και τους υπαλλήλους της Εκτελεστικής Επιτροπής που με βοήθησαν. Ευχαριστώ τους και, και όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν καταθέτοντας τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Μουνής για την τόσο αναλυτική σας παρουσίαση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σάλα Φράγκα που είναι ο σκιώδης εισηγητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Τα έγραψε όλα πάρα πολύ ωραία και ιδιαίτερα λεπτομερώς, αντικατοπτρίζονται όλες οι προκλήσεις οι οποίες ε, ε, έχουν ε, οριστεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εμείς συμφωνούμε γενικότερα με τις αρχές της εισηγήτριας, να αποκαταστήσουμε όλα τα ποσά για την πολιτική γυκνίαση σε ανατολικά και νότια, θεωρούμε πολύ σωστά αυτά που είπε για την Παλαιστίνη, για επίσης για το μέσο της προέναξης, όπως επίσης και για τα άλλα επιχειρήματα που ανέφερε στην αρχή της παρουσίασής της. Δεν είμαστε κατά της αποκατάστασης των πιστώσεων, για τους παρατηρητές εκλογών <coughs> και για την Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων. Εγώ πέρυσι ως εισηγητής αυτής της Επιτροπής ζήτησα να αυξηθούν τα κονδύλια παραπάνω από αυτό το οποίο πρότεινε η Κομισιόν στο προσχέδιο προπολογισμού. Και η Υπηρεσία Εξωτερικών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική με τις προτάσεις αυτού του Κοινοβουλίου. Πέρυσι είχαμε μια κακή εμπειρία. Εγώ είχα την δυνατότητα να τα μεταφέρω όλα αυτά στην κυρία Άστον και είναι λογικό ότι αν το Κοινοβούλιο καταβάλει δημοσιονομικές προσπάθειες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προσπάθειές του. Για το άνοιγμα αντιπροσωπιών στα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Αναφέρθηκε η συγγήτρια και για το άνοιγμα αντιπροσωπεία στο Ιράκ και αυτό βάσει των ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρελθόντος. Εγώ ειλικρινά έχω αμφιβολίες. Για το πώς η ομάδα μου θα δεχτεί ένα άνοιγμα αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη, η συγκυρία και η Αραβική Άνοιξη θα πρέπει να μας ε, κάνουν πιο σόφρονες, ε, πιο συγκρατημένους προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα έπρεπε να αναφερθούμε στα ψηφίσματα τα οποία προηγουμένως έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο αλλά το να είμαστε πια τόσο ανοιχτοί δεν νομίζω ότι με αυτή τη συγκυρία είναι ένα καλό πολιτικό μήνυμα. Τώρα κυρία Πρόεδρε θέλω να σας πω ότι συμφωνούμε με τις τροπολογίες Γκουαλτιέρη για τις εξωτερικές υπηρεσίες της Ένωσης. Δεν καταλαβαίνω γιατί το σχέδιο ψηφίσματος που θα πρέπει να συνοδεύει την ψηφοφορία των ποσών που θα ψηφίσουμε σήμερα το βράδυ δεν θα ακολουθήσει γιατί το ψήφισμα ακολουθεί το σχέδιο. Δεν ξέρω τώρα έλειψε χρόνος. Πάντως μας ενοχλεί εμάς να ε, μας, ε, μας δημιουργεί μια καλή ευκαιρία για να για να κρατήσουμε ε, μία σχετική ευελιξία στη δημοσιονομική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή και τις τρέχουσες εξελίξεις στη Λιβύη. Γενικότερα λοιπόν κυρία Πρόεδρε αυτές είναι οι θεωρήσεις εξ του ΕΛΚ. Συμφωνούμε με τις πιστώσεις πληρωμών που προτείνουν οι φιλελεύθεροι για την διασυνοριακή συνεργασία και το γενικό σχέδιο που μας παρουσιάζει η συγκήτρια είναι ικανοποιητικό και την χάνουμε και θετικών απαντήσεων στα ζητήματα που έθεσε η ομάδα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα για να απαντήσει εν ε, μέρη. Θα το πράξει ήδη κυρία Μινίθ βέβαια. Ε, υπήρξε εδώ ένας διαχωρισμός των θεμάτων γιατί για το σχέδιο γνωμοδότησης έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο, για τις τροπολογίες πρέπει να αποφασίσουμε πολύ σύντομα θα απαντήσει η κυρία Μινής. Αλλά δίνω προηγουμένως το λόγο στην κυρία Γιάχτεμάκη για τη φιλελεύθερη ομάδα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω όλους. Ελπίζω ότι περάσατε καλές διακοπές και είσαστε όλοι δυνατοί και έτοιμοι να εργαστούμε το φινόπωρο. Τα πράγματα ήταν λίγο καλύτερα, ήμασταν πολύ πιεσμένοι στο τέλος του, <clears throat> της προηγούμενης ε, κοινοβουλευτική χρονιά τον Ιούλιο και τον Ιούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Μούνιθ για την πολύ καλή εργασία της. Και εγώ με μεγάλη χαρά θα υποστηρίξω και φυσικά και η πολιτική μου ομάδα μία σειρά από τροπολογίες. Θα ήθελα να σταθώ λοιπόν σε μέσα από αυτές τις τροπολογίες. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες για την Παλαιστίνη. Ελπίζω θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση η οποία θα λάβει υπόψη την ανάγκη να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για την Παλαιστινιακή Αρχή. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες οι οποίες έχουν σαν στόχο να δημιουργηθεί μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράν, εδώ συμφωνώ με τον κύριο Σαλαφράγκα, πρέπει να τονίσω ότι η ομάδα μου δεν έχει τίποτα εναντίον της ιδέας αυτής, αλλά δεν είμαι πεπισμένη ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού είναι ο σωστός τρόπος να προωθήσουμε <clears throat> ένα τέτοιο εγχείρημα, ιδίω σε μια χώρα σαν το Ιράν. Να δημιουργήσουμε λοιπόν μια αντιπροσωπεία στο Ιράν, αυτό είναι ένα σοβαρό πολιτικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και εγώ θα ήθελα εδώ να ακούσω τις απόψεις της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής δράσεις σε σχέση με το θέμα αυτό, εάν είναι κάποιος εδώ παρόν θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε ήδη τώρα τις απόψεις τους. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι σε χαλεπούς καιρούς, όπου δεν έχουμε αρκετούς πόρους στον προϋπολογισμό και σοβεί μια οικονομική κρίση, είναι και καθήκον του Κοινοβουλίου, όσο και του Συμβουλίου, να εξασφαλίσει ότι ο προπολογισμό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αυξηθεί μόνο σε περιορισμένο επίπεδο και θέλω να επιστήσω ιδιαίτερα την προσοχή σας σε ορισμένες γραμμές του προπολογισμού που αφορούν υποστήριξη σε υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες. Από ό,τι κατανοώ, τα κονδύλια εδώ <clears throat> που προβλέπονται βασίζονται στο πολιετές πλαίσιο, αλλά αν η ικανότητα απορρόφησης των χωρών αυτών δεν αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό όπως και η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει σοβαρά να αναθεωρήσουμε τις ε, απόψεις μας σε σχέση με αυτές τις υποχρεώσεις και τις, τα κονδύλια. Οι υποχρεώσεις μας πρέπει να εκπληρούνται, αλλά μπορεί να γίνει αυτό μόνο επί τη βάση των πραγματικών αναγκών. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν και σας ευχαριστώ και πάλι για την πολύ καλή συνεργασία σας. Σας ευχαριστώ, και Πρόεδρος, και ε, Γιέχτε Μαχή. Ο κύριος Αλασί έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την συνάδελφο Μουνής για το έργο της για το σχέδιο προπολογισμού. Όμως θέλω να τονίσω μερικά πράγματα. Το ένα είναι η Παλαιστίνη. Στηρίζω απόλυτα την τρέχουσα πρόβλεψη. Πρέπει να δείξουμε συγκεκριμένη στήριξη και αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Άρα πρέπει να υπάρχει η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί και τα ποσά αυτά να είναι στη διάθεσή μας. Υπογραμμίζω λοιπόν όλος ιδιαίτερος και τονίζω την ανάγκη επειδή η κατάσταση είναι αυτοί που είναι στην περιοχή. Το ίδιο ισχύει και για το Αφγανιστάν. Εγώ υπέβαλα μία τροπολογία με 27 υπογραφές από διάφορες πολιτικές ομάδες. Και αυτό γιατί πολλοί συνάδελφοί μου είπαν να παρουσιάσουμε κάποια συνέχεια με τη νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν. Σε ένα χρόνο έπρεπε να παρουσιάσουμε κάποια αναλλακτική λύση για τη χώρα. Άρα είναι μια δοκιμασία όσον αφορά την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά θα πετύχουμε μόνο αν βρούμε και τα χρήματα να στηρίξουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Είναι πολύ περίεργο λοιπόν να έχουμε μια έκθεση για μια τόσο μεγάλη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην έχει καμία επίπτωση αυτή στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω συνεπώς την ανάγκη που υπάρχει να εγκριθεί η τροπολογία αυτή. Πρόκειται για 50 εκατομμύρια ευρώ για ένα από τα στοιχεία κλειδί της έκθεσης. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, ιδιαίτερα αν το συγκρίνουμε με τον αντίκτυπο που θα έχει το ποσό αυτό συνολικά στην ειρηνευτική διαδικασία και ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν. Συνεπώς ζητάω από τους συναδέρφους να στηρίξουν την τροπολογία αυτή. Στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει αρκετό περιθώριο για αυτή τη μικρή τροποποίηση. Ο προπολογισμό δεν είναι ένα τέλειο μέσο. Έτσι καλώ υπάρχουν ε, πολλά παράλογα πράγματα. Εξακολουθούμε να δίνουμε χρήματα σε πλούσιες χώρες. Εξακολουθούμε να δίνουμε χρήματα σε μη αναγκαίε δραστηριοτητε Οπότε πιστεύω ότι μια προσπάθεια εξορθολογισμού του προπολογισμού και συγκέντρωση του προπολογισμού των χρηκονδυλίων, δηλαδή σε χώρε που έχουν ανάγκη όπω είναι το Αφγανιστάν και η Παλαιστίνη, είναι κάτι αναγκαίο. Γιατί είναι θέμα αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που κρίνεται ανάλογα με τέτοιε αποφάσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ κύριε Ράκη. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκόμες. Οι συνάδελφοι παρακαλώ να είναι πιο σύντομοι, ε, γιατί αρχίζει να πιέζει κάπως ο χρόνος. Παρακαλώ κύριε Γκόμες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Μαρία Μουνής για την έκθεσή της. Όχι, κάνει εξαίρετη δουλειά. Και είναι πολύ πλήρης η παρουσίαση που μόλις μας έκανε. Θέλω να την ευχαριστήσω επίσης που έλαβε υπόψη της κάποιες από τις δικές μου προτάσεις που έχουν να κάνουν με τη σύρρηξη των σωμάτων του ΟΙΕ για παράδειγμα, όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών και των παιδιών. Στηρίζω πάρα πολύ αυτά που είπε για την Παλαιστίνη και για το Ιράν. Βέβαια πιστεύω ότι το να ανοίξουμε το διάλογο με το Ιράν και τα λοιπά είναι πράγματα τα οποία είναι πέρα του προπολογισμού. Δεν θα γίνουν, δεν θα υλοποιηθούν όμως αν δεν υπάρξουν και τα αντίστοιχα κονδύλια. Γι' αυτό και πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν αυτά τα κονδύλια. Αυτό είναι που θα μας επιτρέψει μεταξύ άλλων να προχωρήσουμε. Δεν λέω την εγγύηση για το ότι θα προχωρήσουμε, αλλά αν δεν έχουμε αυτά τα κονδύλια Πρέπει να τα έχουμε γιατί έτσι η κυρία Άστον θα μπορέσει να προχωρήσει. Τέλος, θέλω να υπενθυμίσω αυτό που αναφέρεται στο σημείο 6 της γνωμοδότησης που είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνοχή για την ανάπτυξη. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα τομέα όπου εξακολουθούμε να έχουμε σοβαρά προβλήματα. Η μεγαλύτερη, η περισσότερη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάει στην Αιθιοπία. Κάναμε ακρόαση και με την Αναπτυξιακή Επιτροπή Είχαμε και την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπογραμμίζει ότι τελικά έγινε κατάχρηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν κατάφεραν να πάνε στον πραγματικό προορισμό τους. Αντίθετα φτάσαν σε λάθος χέρια που καταπίσαν ακόμα περισσότερο το λόγο της Αιθιοπίας. Και φάνηκε αυτό και σε μια ταινία που έδειξε το BBC τον Αύγουστο. Ευχαρίστως να στείλω το link σε όλους τους συναδέρφους για να το δείτε κι εσείς πολλοί από εμά δεν θα το είδατε, επειδή ήταν Αύγουστος, αλλά και Human Watch ε, είχε μαρτυρίες. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να τα παραβλέπουμε, γιατί εκεί πηγαίνει το μεγαλύτερο μέρος της αναπτυξιακής μας βοήθεια. Έχουμε στείλει για δεύτερη φορά παρατηρητές για τις εκλογές που δεν κατάφεραν καν να παραδώσουν την έκθεσή τους στις αρχές, γιατί δεν δέχονται την κριτική. Είναι παράδεκτο να κλείνει τα μάτια η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό. Αυτό πρέπει να φανεί στον προπολογισμό αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμες, λέει πρόεδρος. Ο κύριος Βέγκετ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κυρία πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα απλώς να υποστηρίξω την ε, τροπολογία αυτή. Χαίρομαι που έχει υποστηριχθεί από πολλούς συναδέλφους για να συνεχιστεί η οικονομική αρρωγή προς την Παλαιστινική Αρχή και προς την Ούνρα στο επίπεδο που είχαμε ήδη στο παρελθόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ε, τιμωρήσουμε τους Παλαιστίνιους στη Γάζα λόγω του γεγονότος ότι τα δύο τελευταία χρόνια δεν χρησιμοποιήθηκαν <clears throat> τα κονδύλια αυτά λόγω του Ισραηλινού αποκλεισμού, λόγω της ε, αδυναμίας να εφαρμοστούν αυτά τα σχέδια τα οποία υποστήριζε η Ούνρα. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι υποστηρίζω το να υπάρχουν κονδύλια ύψους τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για να, να ξεκινήσουν οι ενέργειες για την ε, βαθμία εξάλληψη της καλλιέργειας οποίου στο Αφγανιστάν μέσα σε ένα πενταετές χρονικό διάστημα. Είναι δύσκολο να είναι κανείς αισιόδοξο σε σχέση με τη στρατιωτική κατάσταση στο Αφγανιστάν, τόσο τον μάλλον σημαντικότερο να υποστηρίξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι καθαρά πολιτικού μη στρατιωτικού χαρακτήρα και το οποίο μπορεί να βοηθήσει τη χώρα αυτή να προχωρήσει προς μια θετική κατεύθυνση. Αυτό ήταν και το νόημα της έκθεσης η οποία υπεστηρίχθη με τόσο μεγάλη πλειοψηφία για τη νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Σας ευχαριστώ κύριε Βέγγερ, ο κύριος Φανόρντεν. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία, θέλω να κάνω καταρχήν ένα γενικό σχόλιο. Είναι πολύ εύκολο να δαπανίσουμε περαιτέρω κονδύλια σε διάφορα εγχειρήματα τα οποία θέλουμε να υποστηρίξουμε. Βρισκόμαστε όμως σε μια στιγμή οικονομικής κρίσης για όλη την Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις μας περικόπτουν δημόσιες δαπάνες δεξιά και αριστερά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει και εμείς να κάνουμε κάποιες εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι να αυξάνουμε τις δαπάνες μας. Επιπλέον, χρειαζόμαστε να θεσπίσουμε και κάποια σειρά προτεραιοτήτων. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η κύρια προτεραιότητά μας είναι η νότια οχθή της Μεσογείου και η εξελίξη στη Βόρεια Αφρική. Εκεί πρέπει να δώσουμε την έμφαση. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν αυτό περιορισμός, να υπάρξουν μειώσεις κονδυλίων και μια σωστή ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε επί τη βάση φιλοδοξιών και ιδεατών. Για το συγκεκριμένο θέμα της Παλαιστίνης. Υπάρχουν κάποιες αρνητικές και ανησυχητικές εξελίξεις στην περιοχή αυτή, μεταξύ των οποίων και η πρόταση να υπάρξει μονομερής ανακήρυξη ανεξαρτησίας και δημιουργίας κράτους από την Παλαιστινιακή Αρχή. Αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Μέχρι τώρα όλοι έχουν συμφωνήσει στο ότι αυτό πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας διαπραγματεύσεων. Ό,τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξαρτάται από τη μη παραβίαση της αρχής της συμπεφωνημένης διαδικασίας ειρήνευσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Φανόρ. Ο κύριος Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ. Σημερίζομαι απόλυτα τη γραμμή της κυρίας Μουνιός. Εγώ θα ήθελα απλώς να αναφέρω τις ε, τροπολογίες μου για τις εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες θέλουν, ε, τίνουν στην ε, αποκατάσταση των ποσών του, σχεδίου, του σχεδίου προϋπολογισμού, διότι αυτές οι περικοπές είναι ακατανόητες και ως προς τη φύση τους. Δηλαδή 8.300.000 περικοπές στις αντιπροσωπείες κάτω δηλαδή από το κατεβαίνουμε μειώνουμε και τον προπολογισμό του 2011 περικοπές ε, για δορυφορικές ε, φωτογραφίσεις ε, και για άλλες δραστηριότητες το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τις εξωτερικές υπηρεσίες και τον προϋπολογισμό τους. Αλλά αυτό θα πρέπει να οδηγεί και τις εξωτερικές υπηρεσίες να εντείνουν το διάλογο με το Κοινοβούλιο, κυρίως μετά από τα, όσα προέκυψαν πέρυσι για τον αριθμό των μονίμων υπαλλήλων της Ένωσης ε, επί του συνόλου του προσωπικού των εξωτερικών υπηρεσιών. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να βάλουμε στο αποθεματικό αυτή την αύξηση που ε, επαναφέρει τον προϋπολογισμό με το σχέδιο του προϋπολογισμού εν αναμονή των απαντήσεων που θα μας δώσουν οι εξωτερικές υπηρεσίες για την ισορροπία μεταξύ υπαλλήλων, δηλαδή ποσοστό ένωσης και άλλων υπαλλήλων. Ο κύριος Έκα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρακαλώ να είναι σύντομος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ήθελα απλώς να πω ότι η Κομισιόν παρουσίασε έναν ισορροπημένο προϋπολογισμό. Σας ευχαριστούμε για όλες τις προτάσεις ε, που υποβάλλατε και που στοχεύουν στην αποκατάσταση των γραμμών που περικόπηκαν. Είναι όμως πολύ δύσκολο να βρούμε στο ε, αιτιολογήσεις στο αποθεματικό Για το διαχωρισμό της γραμμής ε, Παλαιστίνης και Ούρατ, εμείς δεν υποστηρίζουμε <coughs> αυτό το διαχωρισμό, γιατί θα δημιουργήσει προβλήματα τόσο στην εκτέλεση όσο και στην ευελιξία. Ήδη είναι δύσκολο εμείς να εφαρμόσουμε τις διάφορες δράσεις για την Παλαιστίνη και άμα μας αφαιρέσουν ακόμη περισσότερη ευελιξία επιβάλλοντάς μας τεχνητά ορισμένα ποσά ε, θα είναι πολύ δύσκολο για μας ε, να τα διαχειριστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Γκέρον από τις εξωτερικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου καταρχήν ως ε, νέος διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσεως, νέος διευθυντής για τα οικονομικά, να εκφραστώ μόνο επί των διοικητικών σημείων για το προϋπολογισμό του 2012. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη συζήτηση σχετικά με την σύσταση αυτής της νέας υπηρεσίας. Θέλω να ευχαριστήσω επίσημα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων ε, έλαβε υπόψη της με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη γνώμη της εισηγήτριας. Να σας αναφέρω όμως μερικές πολύ γενικές παρατηρήσεις πριν εκφραστώ επί των τροπολογιών των μελών της Επιτροπής. Πρώτη παρατήρηση το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων για το 2012 είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που συντάσσει η υπηρεσία από τη δημιουργία της και βασίζεται στην εις βάθος ανάλυση των πραγματικών αναγκών για τη λειτουργία της. Πρόκειται για έναν διοικητικό προϋπολογισμό, οι διοικητικές δαπάνες είναι υποχρεωτικές και επαναληπτικές. Πρόκειται δηλαδή για τις αμοιβέ, για τα νίκια κλπ. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό ο οποίος ε, έχει μία αύξηση αλλά πολύ μικρή, 27 εκατομμύρια ευρώ ε, επί ενό ε, συνολικού προϋπολογισμού πολύ μεγαλύτερου, είναι όμως ποσά το ουσιαστικά για την έπρεθμη λειτουργία της υπηρεσίας διότι ορισμένες αρμοδιότητες δεν είχαν καλυφθεί προηγουμένως και θα πρέπει να εγγραφούν σε αυτόν τον προπολογισμό. Τέταρτη και τελευταία παρατήρηση, όπως αυτό υπόθηκε από την εισηγήτρια. Οι περικοπές του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, άμα δεν διορθωνόντουσαν, θα δημιουργούσαν δυσκολίες το 2012 για τις εξωτερικές υπηρεσίες, όταν είμαστε δηλαδή σε μια φάση επέκτασης. Για τις τροπολογίες θα ήθελα να πω τα εξής. Η εξωτερική υπηρεσία για ε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων υποστηρίζει τις προτάσεις του κυρίου Γουαλτιέρη για την αποκατάσταση του προπολογισμού στα αρχικά ποσά, χωρίς να <coughs> μπουν στο αποθεματικό. Υποστηρίζει επίσης και την τροπολογία της εισηγήτριας της, της της κυρίας Μπράτνερ και της, του κυρίου Σαλαφράνκα για την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Ειρήνη και να, αρχίσει, να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για την δημιουργία του. Για το θέμα όμως του προσωπικού, η τροπολογία της κυρίας Μπράτνερ Ξέρετε ότι εμείς έχουμε οι υποχρεώσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με το καταστατικό των υπαλλήλων, δηλαδή ε, προαγωγές, ε, μισθολογικές αυξήσεις κλπ. Και κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε πρόβλημα. Για την αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναφέρθηκε από πολλούς ε, βουλευτές Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον και σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων συμμερίζεται την άποψη ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή πρέπει να ενισχυθεί. Για το άνοιγμα μίας αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Ευρωπαϊκά, ε, Αραβικά συγγνώμη, Εμμυράτα θα πρέπει θα πρέπει να το εξετάσουμε μέσα σε μια γενικότερη στρατηγική για την περιοχή και το πλαίσιο είναι αρκετά πολύπλοκο. Δεν μπορεί λοιπόν να ληφθεί μια απόφαση παρά μόνο όταν θα πληρούνται οι πολιτικοί όροι, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα. Η η εκπρόσωπος θα συνεχίσει να εργάζεται για την εφαρμογή για, για, των υποχρεώσεων που, για την εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων που ανέλαβε έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέρα. Η κυρία Μουνής για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους όσοι πήραν το λόγο για τα σχόλιά τους και τη στήριξή τους. Η δουλειά αυτή δεν είναι μόνο δικιά μου δουλειά, έχουν συνεισφέρει πολύ με τις τροπολογίες τους και με τις συζητήσεις που κάναμε πριν εκπονηθεί η έκθεση αυτή. Τα θέματα τα οποία παραμένουν κάπως αμφιλεγόμενα. Για το θέμα του Αφγανιστάν, για παράδειγμα, δεν είναι λίγα τα λεφτά, 50 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσαν να ήταν 70, θα μπορούσαν να ήταν και 40 που ζητάνε η Επιτροπή και το Συμβούλιο, όπως για το 2011. Από την άλλη, δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια τα οποία έχουμε βάλει εμείς σε αυτό το σχέδιο προπολογισμού. Στον προπολογισμό δεν είναι δυνατόν στις γραμμές ε, για συγκεκριμένα προγράμματα να βάζουμε περισσότερες λεπτομέρειες. 50 εκατομμύρια δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πάνε εκεί, γιατί εξαρτάται από τον προγραμματισμό που θα κάνει κάθε χώρα και από τα προγράμματα τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή τελικά με την εκάστοτε χώρα. Θα μπορούσε βέβαια κανείς να το διατυπώσει κάπως διαφορετικά, αλλά αν έχουμε την ε, σιγουριά ότι τα χρήματα θα πάνε στον προορισμό τους, το να μιλάμε για μια τέτοια αύξηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών νομίζω ότι δεν θα βοηθούσε. Δεν πρόκειται να εγκριθεί δηλαδή, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να εγκριθεί ένα τέτοιο ποσό. Οπότε η πρότασή μου είναι να διατηρήσουμε το περιεχόμενο της τροπολογίας, δηλαδή ότι ένα σημαντικό μέρος των κονδυλίων που πάνε στο Αφγανιστάν να πάνε στην αντικατάσταση ε, του οποίου ναι, και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τα κριτήριά μας για τις ε, διάφορες λοιπές γραμμές του προπολογισμού. Τώρα, έρχομαι και στο Ιράν. Ίσως εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα συμβιβασμό. Να αναφερθεί δηλαδή το άνοιγμα αντιπροσωπείας στη γραμμή αυτή για το Ιράν, Ιράκ και Γεμένη. Ε? και στα σχόλια να μιλήσουμε για το άνοιγμα αντιπροσωπιών στις χώρες αυτές όπου το ζητάει το Κοινοβούλιο ή σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμαστεί για να ανοίξουν αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Τέλος πάντων να βρούμε μια διατύπωση η οποία να μιλεί ρητά να μην αναφέρει ρητά μία περίπτωση, αλλά γενικά να αναφέρεται σε αυτό το οποίο έχει εγκρίνει μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το άνοιγμα νέων αντιπροσωπιών. Αν θέλετε, εγώ θα προσπαθήσω να βρω μια συμβαστική διατύπωση και θα σας την στείλω πριν ψηφίσουμε. Τίποτα ρητορικό δεν έχει να πει ο προπολογισμό αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει έλλειψη συνοχή. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει καμιά φορά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημαντικό πολιτικό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας και πρέπει να προσπαθούμε να πετυχαίνουμε τη συνοχή του και να υπάρχει μια ενότητα όσο γίνεται περισσότερο όταν φτάσουμε στο, στην ψηφοφορία. Πρέπει όσο γίνεται περισσότεροι να το στηρίξουν. Γι' αυτό και προσπαθούμε να βρούμε την ε, κατάλληλη διατύπωση, ώστε διατηρώντας τις πολιτικές μας αρχές και επιθυμίες, να πετύχουμε συνένεση από όλους τους ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μινής. Σας υπενθυμίζω ποια είναι η πρόθεσμία για τις τροπολογίες. 7 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Η συζήτηση για τις τροπολογίες σε 8 Σεπτεμβρίου. Μπορούμε να κάνουμε μια διακοπή μερικών λεπτών πριν περάσουμε στο σημείο 7. Η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Σόνισον θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Χρειάζεται λίγος χρόνος για να μπορέσουν να αποχωρήσουν οι μη έχοντες εργασία.